Uh, ladies and gentlemen. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να καλωσορίσουμε την Αυστριακή Προεδρία. Βρισκόμαστε στη, ε, βρισκόμαστε στη 26η μέρα των κινητοποιήσεων ενάντια στη μονομερή επιβολή από τη δίκηση ε, άδικων και μη ισορροπημένων συνθηκών εργασία για του διερμηνεί. Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση λοιπόν να σα ενημερώσουμε πω η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ την προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για την προσοχή σα. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε σε τρία λεπτά με την παρουσίασή σας. Πριν από αυτό, θα ήθελα να σας ε, πω πώς ε, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Όπως ξέρετε, σταματήσαμε στις 12.30. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τώρα αλλά ήταν μετά τις 12.30 χωρίς διερμηνία και με την απουσία ορισμένων συναδέλφων, οι οποίοι αποχώρησαν από την αίθουσα. Καταρχήν, ήρθα σε πληθή με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί είχαμε μια γνωμοδότηση για την υγεία και για τις τεχνολογίες για την Επιτροπή Ένβη ήρθα σε επαφή με την εισηγητρία την κυρία Καμπεσόν Ρουίς και η πρόεδρος της Επιτροπής κυρία Βελέα, και την πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Βελεάν. Είναι πανέτοιμες να λάβουν υπόψη αμέσως τους συμβιβασμούς μας, τους οποίους ψηφίσαμε. Δηλαδή, 90% της γνωμοδότησής μας θα ληφθεί υπόψη αμέσως από την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Τώρα οι υπόλοιποι, το 10% πάνω κάτω, θα ψηφιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα, πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Και μου εξήγησαν αρκεί ο χρόνος για ένα μέρος της γνωμοδότησής μας, για να το λάβουν υπόψη μέσα σε μια εβδομάδα πριν την τελική ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ. Επομένω, όλα καλά. Και ολοκληρώνουμε με συμφωνία, με διερμηνία. Γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι παρέντες εδώ ότι υπάρχει ψηφοφορία στις 3 Σεπτεμβρίου. Και στην ημερήσια διάταξη για τις 3 Σεπτεμβρίου είχαμε ψηφοφορία. Επομένως δεν υπάρχει κάτι καινούριο. To have a voting. Αναμενόταν να έχουμε ψηφοφορία εκείνη τη μέρα, επομένω όλα εντάξει. Κυρία Βίρινγκ. Η κυρία Βίρινγκ που είναι η συγγήτρια αυτής της γνωμοδότησης συμφώνησε για μια τέτοια λύση. Είναι η καλύτερη δυνατή λύση για να ολοκληρώσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου και η ΕΝΒΗ θα λάβει υπόψη όλους τους συμβιβασμούς που θα έχουν ψηφιστεί. Η κυρία Καμπεσονρίς μου είπε μόλις πριν λίγα λεπτά ότι γνωρίζει όλους τους συμβεσμούς της Επιτροπής Βιομηχανίας και είναι έτοιμη να τους λάβει υπόψη. Δεν θα ψηφιστούν, υπερψηφιστούν ίσως ε, όλοι οι συμβασμοί από τους συναδέλφους από την ΕΝΒΗ, είναι προφανές, αλλά θα τους λάβει υπόψη η συγκήτρια. Η δεύτερη γνωμοδότηση αφορούσε την COP24. Εγώ ήμουν ε, ο συντάκτης και ο κύριος Πέτερ Λίζη είναι ο κύριος εισηγητής στην Επιτροπή ΕΝΒΗ και συνήθως η διαδικασία είναι πολύ απλή. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, βάσει της καλής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των Επιτροπών μας, συνήθως υιοθετεί όλες ε, τις τροπολογίες της Ήτρες στην έκθεσή της. Και γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ο συμβιβασμός στην Ήτρα ήταν μόνο μία ψηφοφορία για σήμερα, για τις 12.30. Και οι συμβιβασμοί είχαν υπογραφεί από το ΕΛΚ, από τους σοσιαλιστές, το ECR, το ΑΛΔΕ, τους πράσινους και το EFTD. Δύο πολιτικές ομάδες, το ΙΕΝΕΦ και η ΓΚΟΕ, δεν υπέγραψαν το συμβιβασμό. Αλλά όπως ξέρετε έχουμε συντριπτική πλειοψηφία της Επιτροπής μας να συμφωνεί για αυτή τη γνωμοδότηση. Έτσι λοιπόν η ΕΝΒΗ δεν έχει πρόβλημα να τη λάβει υπόψη αμέσως. Ούτε καν θα περιμένει μέχρι τις 3 Ενάτου. Όμως επισήμως θα ψηφίσουμε και τις δύο γνωμοδοτήσεις στις 3 Σεπτεμβρίου όπως ε, είχε και η προηγούμενη πρότασή μας για τις συνεδρίες της Επιτροπής τότε. Έτσι λοιπόν, Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο συμφωνίας στην Επιτροπή μας και για να έχουμε διερμηνία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, Και για να διαφυλαχθεί και η πολυγλωσία στο Κοινοβούλιο. Έχετε παρατηρήσεις, κύριε Γιάροφ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω. Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες σας να επιλύσετε το πρόβλημα. Νομίζω είναι σαφή τα πράγματα με την COP24. Όμως θέλω να θέσω ένα δυνάμει πρόβλημα σε σχέση με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας. Τι θα γίνει αν η Επιτροπή ΤΡΕ απορρίψει το σύνολο της έκθεσης. Δηλαδή, ενώ η Επιτροπή Ένβη θα λάβει υπόψη του ίδιου υιοθετημένου συμβασμού, αλλά αν η τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης είναι αρνητική. Και επομένω δεν εγκριθεί η γνωμοδότηση στην ΙΤΡΕ. Ενώ οι συμβιβασμοί που έχουν ήδη ψηφιστεί σήμερα θα ληφθούν υπόψη από την ΕΝΒΙ. Αυτό πώς θα το λύσουμε, αν υπάρξει μια τέτοια περίπτωση. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η απάντηση. Δεν μπορώ για να σας τη δώσω τώρα, θα σας απαντήσω αργότερα. Λοιπόν, να καλωσορίσω τώρα την Αυστριακή Προεδρία εκ νέου και να ζητήσω συγγνώμη είχαμε αυτές τις προκαταρκτικές ε, συζητήσεις. Σας, λυπώ, ε, σας ζητώ συγγνώμη, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, περνάμε στην ουσία. Δύο λεπτά να βρω την ημερήσια διάταξη. Ε, λοιπόν, έχουμε την πρώτη επίσκεψη από την Αυστριακή Προεδρία. Έχουμε την επίσκεψη του Μοσπονδιακού Υπουργού Παιδείας Επιστημών και Έρευνας, έρευνα πυρηνικά ζητήματα και επίση θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μάργαρετ Σράμποκ, υπεύθυνη για τη βιομηχανία και το ψηφιακό θεματολόγιο. Είστε υπεύθυνη για τα οικονομικά και τις ψηφιακέ υποθέσεις. Και ο κύριος Χάινς Φάσμαν επίσης είναι εδώ μαζί μας ο Παναδικός Υπουργός Παιδείας Επιστημών και Έρευνα. Χαίρομαι πολύ που μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ε, θέματα, γιατί υπάρχουν στενοί σύνδεσμοι ε, μεταξύ της έρευνας ε, και του ψηφιακού θεματολογίου. Θα έχουμε μια κοινή συζήτηση με τους δύο υπουργού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλος σύνδεσμος μεταξύ των δύο. Στην εποχή της βιομηχανίας και το ψηφιακό θυματολόγιο είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η ΙΤΡΕ. Και συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της πράξης για την κυβερνοασφάλεια, που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, που θα προετοιμαστεί στο μέλλον, το πρόγραμμα της νέας αγοράς για τις επιχειρήσεις, το πρώην πρόγραμμα COSME, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Πολύ σημαντικά ζητήματα λοιπόν. Τώρα από τη σκοπιά της έρευνα και της πυρηνική πολιτικής περιλαμβάνονται τα θέματα, το πρόγραμμα πλαίσιο ε, Horizon Ευρώπη, το, Ευρατόμ, το πρόγραμμα Ευρατόμ Έρευνα και αναπτυξη 2021 2021-2025, καθώς και ο Πυρηνικό αφοπλισμός και η διάθεση αποβλήτων. πολλές νομοθετικές προτάσεις. Θα είναι εδώ στο τραπέζι μας και γι' αυτό έχουμε σημαντική συζήτηση ενωπιών μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, ευχαριστώ και τους δύο υπουργού. Σας ευχαριστώ και που είστε έτοιμοι για συζήτηση. Θα είναι απολύτως καθοριστική η προεδρία σας και για τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε πάρα πολλού φακέλου κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας σα. Και είναι προφανή και δική σα ευθύνη. Και εμεί φυσικά έχουμε ευθύνε. Και η Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ράμποκ για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Σα thank you, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, αγαπητοί ευρωβουλευτές, Συνάδελφε κύριε Φάσμαν, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και χαίρομαι επίσης για την εξαιρετική επικοινωνία ανάμεσα σε εμά και στο Κοινοβούλιο. Η Προεδρία μα είναι ε, μεγάλη χαρά και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε καλή συνεργασία. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να σα παρουσιάσω τι προτεραιότητε τη προεδρία μα στον τομέα του εμπορίου, του Διεθνού εμπορίου με έμφαση κυρίω στη βιομηχανία και την ψηφιοποίηση το θέμα που συζητούμε σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο, διότι η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Διαλύονται παλιές συμμαχίε, εμφανίζονται νέοι εταίροι, υπάρχει τεράστια τεχνολογική πρόοδος, παγκόσμιο ανταγωνισμός και ε, αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μαζί να κάνουμε τα βήματα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει στο μέγιστο το δυναμικό που έχει για τη, στον τομέα της ψηφιακής οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τους ε, τρεις κυριότερους ε, τομείς αυτούς. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας αλλά και κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής και Εστονικής Προεδρίας ασχοληθήκαμε και θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση της βιομηχανίας και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Ε, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών μεταξύ άλλων. Η ψηφιοποίηση επίσης μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας έτσι ώστε να ε, εκβιομηχανίσουμε ξανά την Ευρώπη να ανακτήσει η βιομηχανία της ε, Ευρώπης την δύναμη που είχε στην Αυστρία καταφέραμε να αυξηθούν οι επενδύσεις και να επικεντρωθούν οι επενδύσεις στην Αυστρία. Πήραμε λοιπόν από την Κίνα πολλές επενδύσεις ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ε, ρομποτικής. Επίσης, στη Χαλιβουργία βλέπουμε ότι καταφέραμε στην Αυστρία να προσελκύσουμε ε, την ε, βιομηχανία, να προσελκύσουμε κατασκευές. Πλέον ο Χάλιβας ε, έχει ανακτήσει δυνάμεις. Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα βοηθήσουν δίχως άλλο στην οικονομία. Επίσης, πώς θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη βιομηχανία της Ευρώπης. Ε, καταρχάς πρέπει να σταθούμε στα μοντέλα B2B, business to business, να τεθούν νέες βάσεις, να ε, δημιουργηθεί νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τομέα B2C, ε, βιομηχανή, ε, επιχειρήσεις σε καταναλωτές, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι ε, πρωτοπόρες. Ωστόσο, στην Ευρώπη έχουμε δυνατότητες, έχουμε πολλές ευκαιρίες εάν επικεντρωθούμε στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τον ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα χρειάζονται μέτρα τα οποία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να ε, δρομολογήσουμε με ε, τελικό στόχο την ε, ανάπτυξη της βιομηχανίας. Επίσης, οικολογικός σχεδιασμός, οικοσυστήματα πρέπει να δημιουργηθεί φιλικότερο κλίμα προς τις επιχειρήσεις και εδώ βλέπουμε ότι οι νεόφυτες επιχειρήσεις θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέα οικοσυστήματα επιχειρήσεων. Μαζί λοιπόν με εσάς θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τρόπους μείωσης της γραφειοκρατίας, δημιουργίας ελεύθερου χώρου έτσι ώστε να μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπνεύσουν, να αναπτυχθούν. Θα προσπαθήσουμε επίσης να τονώσουμε την βιομηχανία, την καινοτομία, δίνοντας κίνητρα στις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, ψηφιακή ενιαία αγορά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό τομέα. Ε, κύριε Πρόεδρε, εξάλλου αναφέρατε ήδη πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και για εσά αλλά και για εμάς. Και για τους ε, έξι μήνες ε, που θα διανύσουμε έχουμε μεγάλο έργο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτό το εξάμεινο της Προεδρίας μας να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και γιατί, διότι αυτό θα επιφέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Ευρώπης. Ε, υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία που ε, το δείχνουν εξάλλου. Βλέπουμε ότι θα οι προσπάθειες αυτές θα ε, έχουν όφελος 415 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προτεραιότητες ε, της Προεδρίας μας όμως ξεπερνούν το 2019 σε ορίζοντα. Έχουμε πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και εξισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα ή τις ε, πλατφόρμες ε, επιχειρήσεων, τα οποία είναι δύο θέματα που μας ε, απασχολούν και θα μας απασχολήσουν στην Προεδρία μας, ε, έχουμε αρκετές προτάσεις. Τρίτος βασικός τομέας είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Η έλλειψη καταρτισμένου επαγγελματικού εργατικού δυναμικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή την εποχή. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες από χώρα σε χώρα, γι' αυτό θα δώσουμε βάση στην ε, ε, διπλή, διτή εκπαίδευση. Είναι ένα σύστημα με το οποίο έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην Αυστρία και θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ε, το προωθήσουμε έτσι ώστε οι νέοι να είναι ε, επαρκώς καταρτισμένοι και έτοιμοι να βγουν στην αγορά εργασίας αλλά και να καλύψουν τις ελλείψεις σε καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Αυτό θα, θα γίνει μέσω της ε, έμφασης στις ψηφιακές δεξιότητες μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων, μέσω της ε, χρησιμοποίησης της ε, πλής εκπαίδευσης του διτού εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτι άλλο που αφορά την εμπορική πολιτική και μας αφορά πολύ τόσο εσάς όσο και εμάς ε, στην Προεδρία μας. Πρέπει να βρούμε νέους δρόμους, να δημιουργήσουμε νέες εταιρικές σχέσεις, νέες συνεργασίες ποιοτικέ, οι οποίες θα ε, δρομολογηθούν με διάφορες χώρες όπως η Ιαπωνία για παράδειγμα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την ε, δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ε, Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 600 εκατομμύρια καταναλωτές. Ε, παράγεται το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και τεράστιες ευκαιρίες. Τέλος, πρόθεση της ανταγωνιστικότητας, της ε, καινοτομίας. Η καινοτομία είναι η λέξη κλειδί. Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά. Γι' αυτό λοιπόν θα σταματήσω εδώ και προσβλέπω στην συνεργασία και στην εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά τα θέματα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η επιχειρηματικότητα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ε, Επιτροπή μας και τις αρμοδιότητές της. Καθώς και το ψηφιακό θεματολόγιο. Αναφέρατε και την εκπαίδευση επίσης. Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν είναι ε, μία από τις ε, προτεραιότητες της Επιτροπής μας, είναι ωστόσο κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το πρόγραμμα της ε, Αυστριακής Προεδρίας για την ανεργία των νέων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και το 2013 εγκρίθηκε κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικό σας το Αυστριακό πρόγραμμα πήραμε ως υπόδειγμα αποτελεσματικότητας για να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν που κάνατε πριν από 6-8 χρόνια ήταν εξαιρετική λύση για όλους μας, αλλά και οι εμπορικές συμφωνίες θα μας απασχολήσουν ως καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Από την άλλη όμως, η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, ασχολείται και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, διότι αυτές είναι η ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Και νομίζω πως τώρα μπορούμε να περάσουμε αμέσως στον Υπουργό Χάιντς Φάσμαν, Ομοσπονδιακό Υπουργό Παιδείας, Επιστήμης και Έρευνας καθώς και αρμόδιο για ε, θέματα ερευνητικά, πυρηνικά, για τον ορίζοντα ε, ορίζοντας Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας δώσω το λόγο ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Και εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα ε, κομβικά σημεία της Αυστριακής Προεδρίας που έχουν σχέση με την έρευνα και την καινοτομία. Η πρωταρχική μας προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα είναι αναμφίβολα το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 21 με το πρόγραμμα Horizon Europe. Είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένοι για αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Ιουνίου. Άκουσα ότι στην Επιτροπή ΙΤΡΕ έχετε καθορίσει και ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις. Και εμείς προφανώς έχουμε τις δικές μας φιλοδοξίες. Εάν λοιπόν κατορθώσουμε να επιτύχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για τον κανονισμό Horizon Europe, αυτό θα μας καθιστούσε ιδιαίτερα ευτυχής. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, την οποία κατά κάποιο τρόπο θα αξιολογήσω κιόλας Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα συνολικό προεπλογισμό 100 δις ευρώ που πρότεινε για το πρόγραμμα Horizon Europe. Νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και άλλοι στην Ευρώπη θα επιτιμούσαν μεγαλύτερη πρικοδότηση του προγράμματος. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη και με πολλές άλλες προκλήσεις. Το πρόγραμμα λοιπόν Horizon Europe ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και το κρίνω σε ένα υπεύθυνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το πρόγραμμα Horizon Europe κρίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που αποτελούν συνέχεια. Παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι απολύτω απαραίτητο ε, για την ε, θεμελιώδη έρευνα, τα μέτρα Μαρή Κρουντόσκα ε, όπως επίσης και άλλα μέτρα που έχουν σχέση με τις συνολικές προκλήσει, αλλά και οι τεχνολογίε εχμής όλα αυτά κατά την άποψή μου αποδείχθηκε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πρέπει να συνεχιστούν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν βέβαια και αρκετέ καινοτομίε οι οποίες ε, σίγουρα χρήζουν ιδιαίτερη προσοχής στις διαπραγματεύσεις μας. Μια τέτοια νέα ιδέα είναι η ιδέα των περίφημων αποστολών. Αποστολή, στόχος αν θέλετε με την έννοια ότι μας ενδιαφέρει μια τεράστια βεντάλια που ξεκινάει από τη θεωρητική σύλληψη μέχρι την εφαρμογή. Πολλοί συνάδελφοί μου στο Συμβούλιο χαιρετίζουν αυτή την ιδέα. Νομίζω όμως ότι και στο θέμα αυτό θα πρέπει να αποδώσουμε σημασία στο πώς ακριβώς θα επιλεγούν αυτοί οι στόχοι. Και σε τελική ανάλυση ε, τα αποτελέσματα να είναι αισθητά, να είναι απτά, δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών στην Ευρώπη. Μια άλλη σημαντική κοινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος πλαίσιο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Και εδώ πρέπει να σας πω τελείω ειλικρινά ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και σίγουρα αυτές ε, θα αποτελέσουν αντικείμενο των ε, διαπραγματεύσεών μας κατά τους επόμενους έξι μήνες. Αλλά καταρχήν είμαι θετικά διακείμενο σε αυτό το Συμβούλιο να υπάρχει έρευνα με συγκεκριμένες ε, προεκτάσεις και αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό. Προεκτάσεις, και συγκέντρωση σε περίφημες ε, καινοτομίες, ρηξικέλευτες καινοτομίες, μετά να υπάρχει μεγαλύτερη ενίσχυση των παραπροϊόντων και επίσης ε, και μία ιδιαίτερη στήριξη των καινοτόμων εταιριών οι οποίες ε, προβλέπεται να περάσουν στην επόμενη φάση της ανάπτυξής τους. Αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη του προγράμματος πλαίσιο και υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές πρωτοβουλίες οι οποίες και αυτές θα συμπληρωθούν από το ε, καινοτόμο πρόγραμμα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στον στρατηγικό σχεδιασμό. Στρατηγικό σχεδιασμός είναι ένα νέο στοιχείο στο πρόγραμμα πλαίσιο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως να μην παρουσιάζεται διεξοδικά, αλλά κατανοώ την πρόθεση πίσω από αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή η επιθυμία είναι η διαφάνεια, η μεγαλύτερη ευελιξία, αυτό και σε σχέση με ταχύτατα μεταβελόμενες προϋποθέσεις πλαίσιο. Και αυτό που επιθυμεί κανείς είναι και ένας στρατηγικός σχεδιασμός για το πρόγραμμα πλαίσιο. Όλα αυτά βέβαια τα κατανοώ πάρα πολύ καλά γιατί σήμερα είναι πολύ δύσκολο να αναφερθεί, να αναφερθεί κανείς σε συγκεκριμένα θέματα που θα είναι σημαντικά και το 2020. Όμως, αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο και το πρώτο που θέλω να κάνω είναι στις 17 ε, Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, να συναντηθούμε με τους Υπουργούς Έρευνα στη Βιέννη για να έχουμε έτσι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός. Να αναφέρω και άλλο ένα θέμα που είναι σημαντικό για μένα σε αυτό το πρόγραμμα. Ε, είναι η διεύρυνση των ε, καινοτομιών, η εξάπλωσή τους, αυτό που ενδιαφέρει είναι γενικότερα να ενισχυθεί η Ευρώπη ε, σε αυτό το θέμα και να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στο βορρά που έχει μεγαλύτερη πρόοδο στην έρευνα και στον νότο με φτωχότερη εξέλιξη. Στη τελική ανάλυση όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι να ε, γνωρίζουν και τα κράτη-μέλη ότι οφείλουν να προσφέρουν τη δική του τη συνεισφορά και να μην τα περιμένουν όλα από τις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένα θεματολόγιο σε σχέση με την έρευνα και επ' αυτού του θεματολογίου θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη συνάντησή μας στη Βιέννη. Για να δούμε κατά πόσον έχουμε κατορθώσει, να μπορούμε να κατορθώσουμε, να επιτύχουμε έναν ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο που θα είναι ενωμένος και όχι κατακαιρματισμένος. Για να αποφύγουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, βεβαίως και τα κράτη-μέλη έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πλαίσιο και να στηρίξουμε συγκεκριμένους στόχους. Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα αριστείας, αλλά πρέπει να εκπληρεί και, άλλες, και άλλα καθήκοντα, ερευνητικά και πολιτικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon έχουν ληφθεί, έχει ληφθεί μέρημνα παραδείγματο χάρη για προγράμματα όπως το Sharing Excellence, το να διαδοθεί η αριστεία, η τελειότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα για την Αυστριακή Προεδρία και νομίζω αυτό το υπενήχθην ήδη είναι η περαιτέρω εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου. Για μένα αυτή είναι μια σημαντική υπόθεση το innovation divide δεν είναι ε, ο στόχος, είναι κατ' ουσίαν μια προσπάθεια να ε, σφυριλατηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκός χώρο. Οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες χώρες. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν γενικότερα στον χώρο τη έρευνα και τη καινοτομίας. Εξάλλου, θεωρώ ότι οι επιτυχημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, υπήρξαν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια τέτοια επιτυχημένη προσπάθεια, το Joint Initiative, αυτή την κοινή πρωτοβουλία που αναλάβαμε ή αν θέλετε και την χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων κοινών για τη βιομηχανία και τα πανεπιστήμια. Παράδειγμα, η Σλοβενία. Εκεί είχαμε μια πολύ επιτυχημένη διαρθρωτική μεταχείριση. Τον Νοέμβρη, στις συνεδρίες του Συμβουλίου, θα υιοθετηθούν τα συμπεράσματα για την περαιτέρω εξέλιξη αυτού του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου. Και εκεί θα τεθεί ένα κρίσιμο ερώτημα που επιτύχθηκαν οι στόχοι ε, που ενδεχομένως ε, πρέπει να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο για να βελτιωθεί περαιτέρω ο ερευνητικό χώρος. Ε, μία τρίτη προτεραιότητα που θέλω να θίξω αφορά το θέμα των τομεακών πολιτικών στην έρευνα και επ' αυτού είμαι πεπισμένος ότι οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, τομεακές πολιτικές. Νομίζω η λέξη συνέργεια είναι μια λέξη συχνά χρησιμοποιούμενη, μερικές φορές ε, θεωρείται και μαγική λέξη για, τον, ε, για τη διασύνδεση ε, διαφόρων πολιτικών. Αυτό όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή το θέμα είναι πώς μπορούμε να προσελκύσουμε διαρθρωτικά κονδύλια για να ενισχύσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Η ψηφιακή Ευρώπη, παραδείγματος χάρη. Ε, πώς μπορεί και αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για να στηρίξει την έρευνα και την ε, καινοτομία. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να καταστήσουμε χρήσιμες τις διαφόρων μορφών ε, συνέργειες. High performance computer, συγκεκριμένο άλλο παράδειγμα για το πώς ακριβώς μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί συνέργειες ε, για να υπηρετήσει την έρευνα. Σε τελική ανάλυση, Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Γνωρίζουμε τον προορισμό μας. Ο προορισμός μας είναι μια Ευρώπη με προτεραιότητα την έρευνα και την καινοτομία. Μια Ευρώπη η οποία σε τελική ανάλυση μπορεί να σταθεί επίση όρη στον ανταγωνισμό με την Κίνα και τι ΗΠΑ. Αυτό είναι ο τελικό μα στόχο και χαίρομαι πάρα πολύ που θα διανύσουμε, ελπίζω τουλάχιστον, από κοινού το δρόμο προ τον τελικό στόχο. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργού για τις παρουσιάσεις. Ήταν πολύ σαφείς για μας και σας ευχαριστούμε και για το έργο σας, για τις δραστηριότητές σας και να πω ότι είναι εξαιρετική ιδέα από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια συνεδρίαση για το πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο από σκοπιά χρηματοδότησης μετά τη γεωργία και τη διαθροτική πολιτική. Το τρίτο μεγαλύτερο πρόγραμμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε 7 χρόνια ισχύει μάλλον για 7 χρόνια και είναι τουλάχιστον τρει φορέ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Ε, δεν έχουμε λοιπόν ε, τόσο μεγάλα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω ε, μόνο για του νέου. Έχουμε το εράσμους, είναι το διπλό σε σχέση με το παρελθόν. Όμω έχουμε αυξημένε ευθύνε στα χέρια μας γιατί ξεκινήσαμε από 15-16 εκατομμύρια, τώρα, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, τώρα έχουμε φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Είναι φανταστική η πρόοδος, μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσίασή σας. Να περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Καταρχήν το λόγο θα πάρουν οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων. E Εκ μέρου του ΕΛΚ, η κυρία Πιλάρ Καστίγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. And ορίζω και τους δύο υπουργού που εκπροσωπούν την Αυστρική Προεδρία. Πρέπει να πω ότι ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένη όταν είδα τις τρεις σας προτεραιότητες και πρόσεξα ότι η δεύτερη ήταν ακριβώς η ψηφιοποίηση. Πώς θα καταστήσουμε την οικονομία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική, να μεγεθυνθεί και να δώσει περαιτέρω ευκαιρίες για ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό και συμφωνώ απόλυτα με αυτό είναι μέσω της ψηφιοποίησης. Είναι μια προσέγγιση που μου αρέσει πάρα πολύ. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες συγκεκριμένε πτυχέ όπου μπορείτε να κάνετε κι εσείς κάποια πράγματα στην Προεδρία σας. Ήδη έχουμε ψηφίσει μια σειρά νομοθετικών φακέλων που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ψηφιοποίηση. Ψηφίσαμε την πολιτική συμφωνία, τον ε, κώδικα για τις ε, ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ε, επίσης, ψηφίσαμε και την πολιτική συμφωνία σήμερα, αλλά ψηφίσαμε και για το θέμα της ασφάλειας. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμείς φάκελοι. Ξέρετε όμως ότι η Προεδρία μπορεί να αναλάβει δράση, όχι μόνο γιατί εσείς είστε υπεύθυνοι για να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία σε ένα φάκελο, αλλά γιατί μπορείτε να αρχίσετε να διαμορφώνετε και την θέση του Συμβουλίου σε ένα συγκεκριμένο φάκελο και έτσι δεν γίνει μάλλον όταν θα μιλήσουμε για ειδική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ψηφιακής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στο πρώτο ευρωπαϊκό ψηφιακό πρόγραμμα και προσπαθούμε να έχουμε μία πρικοδότηση, μία επένδυση του στις τάξεις του 9,2 δισεκατομμύρια. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι δεν θα έχουμε τριμερείς διαλόγους στο τέλος της Προεδρίας σας, όμως εσείς τώρα μπορείτε να κάνετε πολλά. Η δική μου ανησυχία και πολλών εξημών είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα 9,2 δισεκατομμύρια. Αυτά καθ' αυτά στον προϋπολογισμό και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο αυτή. Δεν ε, μπορούν ε, κατά κάποιο τρόπο να κατακαιρματιστούν και να δοθούν σε άλλα προγράμματα. Παίρνοντα χάρη στο Horizon ή στις επενδύσεις. Που θα κάνει το Horizon στον τομέα της ε, ψηφιακής έρευνας. Νομίζω ότι το καθένα από τα τρία που έχουμε να είναι ξεχωριστά και να έχουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τα 9,2 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει αυτά να έχουν το δικό τους ε, προσδιορισμό στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτό και αν μπορείτε να οθήσετε ε, το Συμβούλιο προς αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Thank you very much. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Είσαι Βελγίδα. Έχεις ε, συμφωνήσει με το αποτέλεσμα με τον κύριο Μαρτέν. Είναι απαραίτητο να συμφωνήσετε. Γιατί εντός των σοσιαλιστών δεν θέλουμε να έχουμε κανένα big bang, μεγάλη έκρηξη στην πολιτική σας ομάδα. Μην, μην ανησυχείτε, είναι μεταξύ μας. Ισοπαλία θα είναι, μάλιστα. Πέναλτις, λέει ο πρόεδρος. Ξέρετε, δεν έχουν χάσει οι Βέλγοι ούτε έναν αγώνα. Τα κέρδισαν, τους κέρδισαν όλους και δεν πήγαν καν στα πέναλτι. Δεν ξέρω. Κατλίνη, τέλο πάντων, έχει το λόγο. No, Austria my even Spain. Ακόμη και η Ισπανία και η Γερμανία δεν εκπροσωπούνται. Η Πορτογαλία δεν εκπροσωπείται. Κανένας δεν εκπροσωπείται. Αλλά και η κυρία Βιέρινκο. Δύο προ ένα για το Βέλγιο. Εντουάρτ, λυπάμαι, λυπάμαι. Δύο προ ένα το Βέλγιο εδώ στην αίθουσα. Δεν μπορεί να τα καταφέρεις. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα απευθυνθώ σε εσά, γιατί θέλω να σα ε, ρωτήσω μία γενική ερώτηση για τη βιομηχανία και την αυτοβιομηχανία πιο συγκεκριμένα, γιατί νομίζω ότι είναι πήγον το θέμα. Διαφωνήσαμε πολύ σε αυτή την επιτροπή, αλλά νομίζω ότι τείνουμε να συμφωνούμε στο γεγονός ότι χρειάζεται η Ευρώπη ε, μια εύρωστη βιομηχανία που να λειτουργεί καλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε πολλούς ανθρώπους που απασχολούνται σε αυτή τη βιομηχανία και ανησυχώ πολύ γιατί δίνουμε μια μάχη που νομίζω ότι είναι η λάθος μάχη. Είχαμε μια ψηφοφορία σήμερα το πρωί για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυτοκινήτων. Εντάξει, δεν είναι στο δικό σα χαρτοφυλάκιο, αλλά υπάρχει μια πολύ στενή σύνδεση μεταξύ αφενό των φιλοδοξιών που πρέπει να έχουμε για το κλίμα και την ε, ε, καθαρή ατμοσφαιρική και την καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά ε, και σε σχέση με το μέλλον αυτής της βιομηχανίας. Γιατί συχνά μα λείπει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ολιστική προσέγγιση. Έχουμε την νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια φενό και στη συνέχεια έχουμε νομοθεσία που σχετίζεται με την έρευνα και την ανάπτυξη και τέτοια. Πρέπει να τα συνδέσουμε αυτά για να έχουμε ένα όραμα για την αυτοβιομηχανία που θα λαμβάνει υπόψη και το μέλλον. Και Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πετύχουμε φιλόδοξου στόχου για το δεξίδιο του άνθρακα και τι εκπομπέ και είναι απαραίτητο γιατί θα αρχίσουν διαφορετικά καταναλωτέ να αγοράζουν ιαπωνικά και κινέζικα αυτοκίνητα. Όμω, ένα θέμα που σχετίζεται συχνά είναι η έρευνα και η ανάπτυξη και η στήριξη αυτών και οι επενδύσει στι υποδομέ. Και αυτή είναι η ερώτησή μου, γιατί αυτό είναι εντό του δικού σα χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, θα αναπτύξουμε μια νέα επενδυτική πολιτική, ένα νέο επενδυτικό εργαλείο, το U-Invest, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε μία λίστα προτεραιοτήτων ότι θα ε, επενδύσουμε σε συγκεκριμένες υποδομές και υποδομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το ένα. Δηλαδή αυτό που λέμε περί του αυγού και της κότας. Ε, Κανένα δεν θα αγοράσει τα αυτοκίνητα αν δεν υπάρχει υποδομή. Όμω είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά τα κρατήματα δεν ε, αναλαμβάνουν δράση. Αυτή είναι η εκκλησία μου και η ερώτησή μου προ τα εσά. Πώ μπορούμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και να συσχετίσετε με τη φιλόδοξη νομοθεσία για τι εκπομπέ διεξουδίου του άνθρακα, τι επενδύσει στι υποδομέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αγοράσουν οι άνθρωποι αυτά τα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα οδηγήσουν βεβαίως και να υποστηρίξουμε και την έρευνα και την ανάπτυξη. Και τελευταία ερώτηση. Δεν ε, ξέρω πώς σχετίζεται αυτό με την ενέργεια περισσότερο. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή τη βιομηχανία έχουν ε, τα κατάλληλα προσόντα και τις δεξιότητες για να ασκήσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κασνοντέμσκι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση στους κυρίους υπουργού. Θέλετε να μιλήσω γερμανικά? Υπάρχουν δύο πράγματα που πολλές φορές ε, παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη και σχετίζονται πολύ με το ψηφιακό ζήτημα και με το θέμα της βιομηχανίας και της ενέργειας. Είναι σημαντικό να ασχοληθεί η Αυστρική Προεδρία με αυτά τα θέματα. Αφενός, έχουμε το θέμα των δικαιωμάτων δημιουργού στην ψηφιακή εποχή, σε αυτό το ψηφιακό χώρο. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται για το θέμα αυτό για να δούμε ποια θα είναι τελικά η θέση του Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του δημιουργού. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο δεν έχουν ξεπεραστεί συγκεκριμένα εμπόδια, δηλαδή πώς θα διασφαλίσουμε την ελευθερία στο διαδίκτυο και τα συμφέροντα των χρηστών. Μας έχουν στείλει πάρα πολλά email τους τελευταίους μήνες αφενό και αφετέρου πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, ευρωπαϊκή δημιουργική βιομηχανία, του Ευρωπαίου δημιουργού. Τι θα συμβεί στο Συμβούλιο, θα ήθελα να μου πείτε κάτι, ό,τι μπορείτε να μου πείτε και ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και να έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο για το θέμα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω. Η δεύτερη είναι κάτι τελείως διαφορετικό όμως επίσης φτάνει στην κοινή γνώμη. Και έχει γεωπολιτική σημασία. Έχει να κάνει με την αναθεώρηση της οδηγίας του αερίου. Γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο εδώ και οκτώ μήνες δεν μπορεί να φτάσει σε κοινή θέση για να ξεκινήσουν ε, αυτές οι συζητήσεις, αυτή οι τριμερείς διάλογοι. Όμως η ανανέωση αυτής της οδηγίας αφορά ε, ένα πολύ επίμαχο σχέδιο, το Nord Stream 2. Ένα, σε ένα γερμανικό Ινστιτούτο, στην τελευταία εκδοσή του, τον ε, Ιούλιο, μας είπε ότι από οικονομική σκοπιά αυτό το έργο δεν έχει κάποιο νόημα. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα, κύριοι, να σας ρωτήσω τα εξής στο Κις μέλλον η Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα στην Κορεπέρ. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η Αυστριακή Προεδρία είναι ρητορική βέβαια, έτσι, με κατανοείτε, είναι ρητορική ερώτηση. Μπορεί να είστε ουδέτεροι και να πόσχετε από το γεγονός ότι αυτή η αυστριακή εταιρεία που είναι στο consortium συμμετέχει εκεί. Όμως, έχω ακόμα δύο ερωτήσεις. Ο κύριος Υπουργό υπενθύμησε το πρόγραμμα του Horizon Europe και την τεράστια δυναμική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα μπορούσαμε να καταστήσουμε δυνατόν έτσι ώστε η σημερινή Μαρή να μην, ε, Μαρία Σκοντόφσκα μάλλον να μην χρειάζεται να πάει στη Γαλλία και να γίνει η Μαρή Κιουρί Υπάρχει μια σειρά δηλαδή ταλέντων και στη Βαρσοβία και σε άλλες πολωνικές πόλεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να μετακινηθούν. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Λίνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία και κύριε Υπουργέ, για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις σας. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για την έμφαση που δώσατε στην ψηφιοποίηση στο πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό σημάδι. Κυρία Υπουργέ, μας παρουσιάσατε το όραμά σας ή να το πω διαφορετικά την οπτική σας ε, γωνία ή την ε, οπτική γωνία της Αυστρίας για το θέμα αυτό και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ε, η συνάδελφος Καστίγιο Βέρη. Είμαι συνσηγήτρια της έκθεση στην οποία ανέφερε η κυρία Καστίγιο και νομίζω πως έχουμε καλύψει πολλά θέματα στην έκθεσή μας από αυτά που αναφέρατε, δηλαδή το υπολογιστικό νέφος, ψηφιακές δεξιότητες κτλ. Ελπίζω λοιπόν η, η Αυστριακή Προεδρία να ε, ακολουθήσει και ίδια αυτές τις ε, προτεραιότητες έτσι ώστε να επιταχύνει τη διαδικασία και να δρομολογηθεί ε, το θέμα αυτό. Μετά, στο θέμα της έρευνας, ελπίζω και εσείς να καταφέρετε να έχουμε θετικά αποτελέσματα ε, και επιτυχία στον τομέα αυτών. Η ψηφιοποίηση έχει μεν παρουσιαστεί ως προτεραιότητα, όμως θα με ενδιέφερε να μάθω ακριβώς πώς θα το χειριστείτε. Ποια είναι τα ε, κεντρικά σημεία που θα δώσετε έμφαση. Στην παρουσίασή σας μας δώσατε την ε, αυστριακή προοπτική, ε, ως αυστριακή υπουργό φυσικά, αλλά θα θέλαμε όμως να μας αναφέρετε και το όραμα της Αυστριακής Προεδρίας για την Ευρώπη, για το πώς η Ευρώπη θα ηγηθεί στον τομέα της ψηφιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάβορ, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μια ερώτηση προς τον Υπουργό Φάσμαν δεδομένου ότι είστε επίσης αρμόδιος και για πυρηνικά ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο θέμα της συνθήκης Ευρατόμ. Η συνθήκη αυτή είναι 60 ε, ετών, ε, είναι, μια συνθήκη που δεν έχει ε, τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 60 χρόνια και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η ενεργειακή αγορά είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα όταν υπεγράφει η συνθήκη Ευρατόμ είναι λίγο πολύ λοιπόν παροχημένη και νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να δούμε πώς θα μεταρρυθμιστεί. Η συνθήκη αυτή επίσης έρχεται σε αντίφαση με άλλους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ε, όσον αφορά τις δημόσιες ε, συμβάσεις. Να σας υπενθυμίσω πως υπάρχουν και προσφυγές τις οποίες έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση της Αυστρίας για ε, ένα πυρηνικό εργοστάσιο στα σύνορα ε, με την Ουγγαρία. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ε, συνθήκης Ευρατόμ και το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα τη συνθήκη αυτή και τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως έχετε ευκαιρία να βελτιώσετε και να εναρμονίσετε τη νομοθεσία έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις υπόλοιπες ε, συνθήκες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν η κυβέρνησή σας είναι έτοιμη να ασχοληθεί με αυτό το θέμα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους τώρα της ομάδας inf e ως συνήθως η κυρία Κάπελ. Είστε εκπρόσωπος της ΕΝΕΦ σε πολλούς τομείς. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ε, μιλώ πριν από τους άλλους, από δύο συντονιστές, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, κυρία Σράμποκ, κύριε Φάσμαν, που ήρθατε σήμερα και για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Ε, καταρχάς αναφερθήκατε στην ενίσχυση της βιομηχανικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσυπογράφουμε, συμφωνούμε απόλυτα ε, με το όραμα για την Ευρώπη του 2020. 20% επιπλέον ψηφιοποίηση. Η Αυστρία, όπως και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπολείπονται ακόμα, έχουν πολύ δρόμο να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, χρειάζεται ε, να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Ακριβώς επειδή η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της παγκοσμίω. Η ψηφιοποίηση είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η στρατηγική ψηφιοποίηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ε, αναφερθήκαμε στο πρόγραμμα του Digital Europe με το οποίο καθίσταται σαφές ότι η ψηφιοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό, το οποίο μας το είπατε κι εσεί εξάλλου. Ε, υπάρχει δυναμικό αύξηση, το είπα κατά 15 δισεκατομμύρια ανά έτος. Επίσης, αναφερθήκατε στις ψηφιακέ δεξιότητες. Το πρωί στην Επιτροπή ψηφίσαμε μία έκθεση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται άμεσα με την ψηφιοποίηση. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου στο μέλος. μέλλον. Γι' αυτό και για εμάς και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πολύ σημαντική και ε, φυσικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και οι οργανισμοί που ασχολούνται με αυτό. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα ενιαίας πιστοποίησης. Γι' αυτό λοιπόν εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό, πώς θα φροντίσετε έτσι ώστε να συγκλίνει η νομοθεσία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει διαφορετική νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Έπειτα, Βρισκόμαστε σε απρόβλεπτους καιρούς, το είπαμε και εμείς, υπάρχουν διάφορες διεθνείς συμφωνίες με την Αυστραλία, με την Νέα Ζηλανδία για παράδειγμα που βρίσκονται σε καλό δρόμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει όμως να δούμε τις εμπορικές συμφωνίες στο συνολικότερο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε με αυτές και την ψηφιοποίηση έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση της Ευρώπης και η βιομηχανία της Ευρώπης. Επίσης, ε, προς τον κύριο Φάσμα να αναφερθήκατε στον ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα αυτό. Ακούσατε και από τους ε, συναδέλφους ε, σχετικές ερωτήσεις και δίχως αμφιβολία θα είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φυσικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις οικονομικές προβλέψεις. Θέλουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα, να χρηματοδοτηθεί περισσότερο η έρευνα και η ανάπτυξη, διότι αυτές είναι η κινητήριος δύναμη για την Ευρώπη. Θα οδηγήσουν σε επενδύσεις, θα οδηγήσουν σε αύξηση τη ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι η δική σα θέση για την αύξηση ε, της χρηματοδότησης του ορίζοντα Ευρώπη στα πλαίσια του επόμενου ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα γίνει από τα διαρθρωτικά ταμεία, με κάποιον άλλο τρόπο, ε, πώς θα συνδέεται με αλλού επί παράδειγμα, με την ε, Γεωργία. Επίσης, υπάρχουν ε, σημεία τα οποία βελτιώνουν το πρόγραμμα, το μέλλον του Ορίζοντας Ευρώπη. Το θεωρούμε πολύ θετικό. Αναφερθήκατε επίσης στην, ε, στις αποστολές και στην, αποστο, και στην αποστολή σας, το έργο σας, ε, ότι θεωρείτε προσωπική σας αποστολή να μειωθούν τα, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρώ πως έχουμε κοινού στόχους και πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να συνδεθεί αυτό με τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την άποψή σας και τη θέση σας ε, της Προεδρίας δηλαδή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος ε, των ερωτήσεων από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και τώρα θα περάσουμε σε ερωτήσεις από άλλους συναδέλφους. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να είστε σύντομοι και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρούμπιγκ. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους δύο υπουργούς, γιατί βεβαίως στην Ευρώπη υπάρχει ένας ενθουσιασμός, όχι μόνο λόγω της Αυστριακής Προεδρίας, αλλά κυρίως ε, διότι θα καθοριστεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα 7 χρόνια. Και ως εκ τούτου θα εντοπιστούν και νέες προτεραιότητες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την πολιτική μας, έτσι ώστε να την εστιάσουμε περισσότερο στους πολίτες. Σήμερα μιλήσαμε για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ε, και εκεί ε, είπαμε ότι οι τιμές ε, για την επικοινωνία θα πρέπει να προσανατολίζονται και στο κόστος. Σε διεθνές επίπεδο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Στην Ευρώπη ένα gigabyte κοστίζει περίπου 7 ευρώ. Σε άλλες υπήρους, αν θέλει κανείς ε, να το χρησιμοποιήσει αυτό το 1 gigabyte μπορεί να φτάσει και στις 19.500 ευρώ. Αυτό αφενός έχει σχέση με την εμπορική πολιτική, αφετέρου δε και με την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Ε, θα με ενδιαφέρε πολύ να μάθω την άποψή σας από αυτού. Μία ερώτηση για τον κύριο Φάσμαν. Έχουμε τώρα τους ε, υπερυπολογιστές. Εκεί έχει προσχωρήσει και η Αυστρία. Quantum computing. Έχετε προσχωρήσει σε αυτό. Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι σε αυτά θέλουμε να σημειώσουμε πρώτο. Στον προϋπολογισμό ε, τραβήξαμε κόκκινη γραμμή στα 120 δις. Ε, βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει 160 δις ως εκ τούτου με αυτά που επέρχονται έχουμε μεγάλες ευκαιρίες ε, να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία προς όφελος της Ευρώπης. Ο κύριος Νταλούντε. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Φάσμαν για το Horizon Europe. Καταρχήν για την κλιματική δράση. Αν δούμε τον έλεγχο που έγινε για το Horizon 2020, δεν έχει υλοποιηθεί για την περίοδο αυτή ε, λόγω επαρκούς χρηματοδότηση. Ο στόχος ήταν 35%, αλλά βλέπουμε τώρα μόνο 30%. Επίσης, ε, ο έλεγχος αμφισβήτησε αν και το 30% ήταν ακριβές γιατί ε, μπορεί να έχει τον τίτλο κλιματική δράση αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Εσείς ποιες ασφαλιστικές δεκλίδες ε, θα βάλετε για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε το στόχο του 30% στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση. Η διακήρυξη της Βαρκελόνης λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τι δαπάνε για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ του. Είμαστε αρκετά μακριά από το στόχο αυτό. Τι προτείνετε για να πληρωθεί αυτό το κενό και να υπάρξει μεγαλύτερο δυναμικό καινοτομία στην Ευρώπη. Χρονοδιάγραμμα τώρα για το Horizon Europol, εκτό ε, από το Συμβούλιο, βιάζονται να πετύχουν τι προθεσμίε. Αλλά γιατί εμεί να βιαζόμαστε αν το Συμβούλιο δεν έχει καμία διάθεση να το λήξει αυτό γρήγορα. Πώ θα διασφαλίσετε ότι θα πετύχουμε συμφωνία έτσι ώστε να δούμε πρόσκληση υποβολή προτάσεων το 2021. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση προς τον καθηγητή κύριο ε, Φάσμαν. Συνάδελφε, είπατε βέβαια ε, έτσι με κάποιες επιφυλάξεις παρουσιάσατε το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Παραμένει όμως το γεγονός ότι το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ε, θα απομακρυνθεί από το στόχο του 3% γιατί αυτό καθορίστηκε από τους ίδιους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και αν το επιμερίσουμε σημαίνει το ευρωπαϊκό η ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι 97 δις και το υπόλοιπο ανήκει στο 3% στη βιομηχανία και σε όλους τους άλλους φορείς. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι αυτά τα 100 εκατομμύρια πρέπει κανείς να τα εξετάσει με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Μάλλον είναι 100 δις ε, νοσομιλητής. Ε, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχουν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, αν δώσουμε 10 δις για τη Γεωργία, 3,5 δις πηγαίνουν για ένα ε, χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί από τα ερευνητικά κονδύλια. Αν θέλετε δηλαδή, το πρόγραμμα αυτό ε, δεν είναι ικανοποιητικά πρικοδοτημένο. Και ερωτώ, το Συμβούλιο θα απομακρυνθεί από το στόχο του 3%. Και δεύτερο ερώτημα, όσον αφορά στη διαδικασία. Σε πάρα πολλά από τα ερωτήματα που τέθησαν, το Συμβούλιο ήταν εκείνο που είχε δυσκολίες. Το Κοινοβούλιο είχε προτείνει συνέργειες ε, και μετά το Συμβούλιο είχε σταματήσει, νομίζω για τρεις μήνες περίπου, γιατί δεν μπόρεσε να συμφωνήσει στην τελευταία θέση. Εσείς το στόχο του Κοινοβουλίου τον χαρακτηρίσατε φιλόδοξο, αλλά ένας λόγος αυτής της φιλοδοξίας είναι ότι σε αντίθεση με την τελευταία φορά θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στο Συμβούλιο να αναπτύξει ταχύτερα την διαπραγματευτική του θέση. Ε, για δύο μήνες όπως σας είπα υπήρχε μία αναστολή γιατί το Συμβούλιο ήθελε να αφομοιώσει κάποια θέματα και γι' αυτό πέρα από τις δικές μας ε, φιλοδοξίες ποιες είναι όλες οι υπόλοιπες φιλοδοξίες όσον αφορά όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα αλλά και για το να υπάρξουν συγκεκριμένες θέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων. Ευχαριστούμε κύριο Ζωρίνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργή. Καταρχήν, μία από τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας είναι η ψηφιοποίηση. Σε ένα πλαίσιο ότι η ιδέα κλειδί είναι η Ευρώπη που προστατεύει. Το θέμα είναι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιοποίηση για να προστατεύσουμε Δηλαδή, για να συμπεριλάβουμε προστασία, ασφάλεια, την ε, συμπερίληψη και την πρόσβαση. Εγώ είμαι και σκιώδης εισηγητής ε, για τα ψηφιακά και θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Όμως θέλω να θέσω μια μέση ερώτηση γιατί πιστεύω ότι το πώς ε, θα επιληθεί όλο αυτό θα διαμορφώσει και τι θα ακολουθήσει έχουμε μια πρωτοβουλία που ελήφθη από τον κύριο Γιούνκερ, το Wi-Fi for You. Ήταν ε, ουσιαστικά μια ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17.000 υποψηφιότητες είχαμε, από τις οποίες 11.000 υποψηφιότητες εγκρίθηκαν. Και ουσιαστικά από τη Βουλγαρική Προεδρία θα κληρονομήσετε αυτό το ζήτημα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε κύριε Υπουργέ, Ποια θα είναι η δική σας υποστήριξη έτσι ώστε η ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabyte να συμπεριλάβει όλους τους Ευρωπαίους είτε ζουν στις πόλεις, είτε στην Ήποθρο, είτε σε ορεινές ή σε παραθαλάσσιες περιοχές. Και ποιο είναι το όραμά σας, πώς από αυτή την πρωτοβουλία του Wi-Fi for You που ε, χρηματοδοτείται μπορούμε να προσφέρουμε ε, παιδεία, ολοκλήρωση ανάπτυξη, να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να δημιουργήσουμε μια μελλοντική ψηφιακή ταυτότητα. Ουσιαστικά, εγώ πιστεύω για τους καλούς λόγους να μπορέσετε να τα εκμεταλλευτείτε αυτά ως Προεδρία. Κύριε Υπουργέ, ε, είπατε ότι είστε υπουργό ενέργεια, αλλά δεν μιλήσατε για ενέργεια. Ε, Εμεί σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας ψηφίσαμε τις ε, συμφωνίες για την ε, διακήρυξη, τη διακυβέρνηση ενέργειας για την ενεργειακή αποδοτικότητα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μας δώσουν τα πρώτα σχέδια για το 2020-2030, καθώς και τα σχέδια τα μακροπρόθεσμα μέχρι το 2050. Πώ μπορούμε να βασιστούμε στην Αυστρική Προεδρία ότι θα προωθήσετε αυτό το πολύ σημαντικό σχέδιο και την πολύ σημαντική δεσμή μέτρων για την ενέργεια. Ευχαριστούμε. Πιθανότατα είχαμε τη συζήτηση για την ενέργεια, αλλά εγώ δεν είχα πολωνική διερμηνία. Να τα πω και στα αγγλικά αν προτιμάτε. Όχι. Μου είπε όμως η γραμματεία ότι μίλησατε για ενέργεια. Θα πρέπει να θυμάστε ότι το επόμενο θέμα της για διαταξής μας θα είναι μια συζήτηση για την ε, ενέργεια με τον Ελληνικό Υπουργό. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα θέματα ενέργειας σε 20 λεπτά περίπου. Επομένως, ε, θα μπορούσαμε να τα θέσουμε αυτά τα θέματα 20 λεπτά αργότερα. Αλλά θέλετε τώρα να τα πείτε γιατί είναι ο υπουργό μας. Είμαστε κανένα πρόβλημα. Αν κατάλαβα και τι είπατε βέβαια. Και τώρα να πάμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Σαουντάρκας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Αυστριακή Προεδρία για μια ολιστική προσέγγιση. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, στα βιομηχανικά σχέδια έχουμε μακροπρόθεσμες τάσεις και μερικές φορές είναι εύκολο να κάνουμε κάποιες προγνώσεις. Φυσικά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και 50 χρόνια ιστορίας. Αλλά τι έγινε πρόσφατα, στα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε μια τρομερή επιτυχία, ρεξικέλευτες εξελίξεις λόγω των ικανοτήτων των ε, υπολογιστών και των μεγάλων δεδομένων, των μαζικών δεδομένων. Η βιομηχανία αντέδρασε γρήγορα, αυξάνονται εκθετικά οι επενδύσεις και ίσως να παραβλέψουμε κάτι. Στην Ευρώπη είχαμε την ανακοίνωση της Κομισιόν και ξέρουμε ότι στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πολιτικές αντιδράσεις. Τι σκοπεύει ακριβώς να κάνει η Προεδρία, σκοπεύει να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση ή θα ακολουθει την πεπατημένη. Thank you very much, um, Next Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για την Υπουργό. Η πρώτη ερώτηση αφορά την Ευρώπη που προστατεύει γιατί έχετε αυτό το σλόγγαν που αφορά τη μετανάστευση, αλλά έχετε και συγκεκριμένη προσέγγιση, γιατί μου φαίνεται κάπως αφηρημένο το πρόγραμμα. Σε σχέση με την προστασία των θέσεων εργασία, αν η Ευρώπη προστατεύει και τι θέσει εργασία και σας θέτω αυτήν την ερώτηση γιατί έχω και πρακτικό παράδειγμα. Στις 11 Απριλίου έλαβα μια επιστολή σε σχέση ε, με, τον όμιλο από την Αυστρία, την ε, Υπομπάνκ, σε σχέση ε, με την απώλεια θέσεων εργασίας και σε αυτή την επιστολή δεν λάβαμε ποτέ απάντηση. Πώς σκέφτεστε λοιπόν να απαντήσετε, να δώσετε απαντήσεις στην Ευρώπη, αν δεν μπορείτε καν να απαντήσετε σε μια επιστολή. Πέρα ότι είναι δυσάρεστο να μην απαντά κανείς. Το δεύτερο αφορά την έρευνα και τους υπερυπολογισμούς. Για τον κύριο Φάσμαν, την ανταγωνιστικότητα με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα όταν έχουμε ένα τεχνολογικό χάσμα, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές εφαρμογές. Πώς σκοπεύετε να καλύψετε αυτό το χάσμα. Ευχαριστώ. Και τέλος, η κυρία Βίριν. Και να σας ενημερώσω ότι η κυρία Καμπεσόν Ρουίς είναι έτοιμη να δεχτεί όλες τις συμβιβαστικέ τροπολογίες σας με ενημέρωση ότι γνωρίζει τις συμβασικές απολογίες κάθε επιτροπής και είναι έτοιμη να τις δεχτεί. Της είπα λοιπόν ότι κατά 90% έχουμε ψηφίσει την γνωμοδότηση, οπότε πρέπει να τη λάβει πολύ στα σοβαρά. Πριν από μία ώρα συζήτησα μαζί της το θέμα αυτό. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία και κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τον ε, ορίζοντα Ευρώπη. Το Συμβούλιο πράγματι έχει σκοπό να διαπραγματευτεί μαζί μας μέχρι το τέλος της ε, θητείας. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στην νομοθεσία, τα προγράμματα, το ΣΕΦ, ε, τη συνοχή κτλ. Τέλος, προσπαθούμε να βελτιώσουμε μέσω των επενδύσεων την κατάσταση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δίνουμε έμφαση σε αυτό παρά να αποδυναμώνουμε την έννοια της αριστείας και να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Ποια είναι λοιπόν η θέση του Συμβουλίου και της Προεδρίας σχετικά με τη χρήση των ε, διαρθρωτικών ε, ταμείων για να στηρίξουν ε, εθνικούς στόχους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να προτείνω να περάσουμε στο, στις απαντήσεις και θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Σράμπακ έτσι ώστε να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Φάσμαν. Έχετε το λόγο, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συνεισφορά σας και για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, απαντήσω αμέσως Αρχικά από το θέμα της ε, ψηφιακής Ευρώπης, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Η Αυστριακή Προεδρία καλωσορίζει την πρόταση για το Digital Europe για το διάστημα 2021-2027 κατάσταση στην Ευρώπη αλλάζει διαρκώς, όλο ένα και ψηφιοποιείται. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστούμε και εμείς αναλόγως και γι' αυτό χρειάζονται και αντίστοιχε επενδύσει. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς και συμφωνούμε μαζί σας. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό, καθώς και ε, στους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, την ε, κυβερνασφάλεια, την ε, τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την εισαγωγή βέλτιστης της χρήσης ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα, όπως αναφέρατε κι εσείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προηγμένες ψηφιακές ε, δεξιότητες είναι ένα από τα ε, θέματα στα οποία θα δώσει έμφαση η Προεδρία μας. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πως υπάρχουν μελέτες ε, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των πολιτών της Ευρώπης έχει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Φυσικά αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με την απασχόληση και με τις μελλοντικέ θέσεις απασχόλησης, διότι αυτά είναι αλληλένδετα. Επίσης, χρηματοδότηση ε, και το αντίστοιχο πλαίσιο. Να πω εν συντομία ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να το δούμε ως ένα σύνολο. Ε, το Συμβούλιο λοιπόν στα πλαίσια της δουλειά του για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο εργάζεται σε επίπεδο υπουργών. Στις 14 ε, Μαΐου είχαμε την τελευταία σχετική συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών και εμείς συνεχίζουμε από τον προκάτοχό μας με έμφαση στην ψηφιοποίηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ένωση. Η Ενίσα ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής και Εστονικής Προεδρίας και ε, στις 8 Ιουνίου έλαβε χώρα τελευταία συνάντηση όπου και ε, συζητήθηκε ο κανονισμός για τον ε, Ενίσα. Τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχεια και θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό, διότι θέλουμε να προχωρήσει το θέμα. Είναι όμως σημαντικό να πούμε ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για ε, εμάς είναι κάτι που αφορά πάρα πολλούς τομείς. Ε, είναι, έχει ευρύτατη εφαρμογή από τις ψηφιακές δεξιότητες, την καινοτομία και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χρειάζεται να δημιουργηθούν κόμβοι Γι' αυτό για μας ε, είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη όχι μόνο για την Αυστριακή Προεδρία, αλλά για την Ευρώπη γενικότερα, για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφάλεια, ωστόσο, είναι εθνική αρμοδιότητα. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη και να στηρίζουμε ε, τις, ε, τα κράτη-μέλη. Η Αυστριακή Προεδρία θα έχει ρόλο διαμεσολαβητή. Δεν πρέπει βέβαια να ε, αφήσουμε την ευθύνη μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά χρειάζεται καλή συνεργασία και σωστές επενδύσεις. Τέλος, ε, θα ήθελα να σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο αναφέρατε και ε, ορισμένοι από εσά για το πώς δηλαδή θα καταφέρουμε να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις μικρομεσαίες βιομηχανίες και επίσης η Οι πληροφορίες ε, του δημόσιου τομέα είναι επίσης σημαντικό ε, τομέα για εμάς. Χρειάζεται παρκής πληροφόρηση. Βέβαια, νομίζω ότι και ο κύριος Φάσμαν είναι αρμόδιος για να σας πει περισσότερα, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι και ο συναδελφός μου και εγώ ε, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για τη βιομηχανία, να πω εδώ πως ε, θέλουμε να δρομολογήσουμε ένα φιλόδοξο έργο, δηλαδή νέα βιομηχανική πολιτική. Ελπίζουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμη η πρότασή μας. Ε, προβλέπουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης στα πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής που έχει στόχο την, ε, ε, τους ίσους όρους ανταγωνισμού, την προστασία της βιωσιμότητας, όμως και να μην ξεχνάμε ότι στο κέντρο των προσπαθειών μας πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω θα μας βοηθήσουν στο να ε, δημιουργήσουμε δουλειές για τους πολίτες της Ευρώπης. Στην Προεδρία μας έχουμε αυτούς τους ε, τρεις κύριους θεματικούς άξονες, δηλαδή η Ευρώπη που προστατεύει, ε, τον δεύτερο θεματικό άξονα που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση που θα αποτελέσει βάση για ευημερία και ανταγωνιστικότητα. Και εδώ ε, είμαστε έτοιμοι και έχουμε προτάσεις για την προστασία των εργαζομένων. Θέλουμε να προστατεύσουμε και να, ε, να προστατεύσουμε τις ε, θέσεις απασχόλησης Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες ικανότητες έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της αγοράς σε δεξιότητες. Επίσης, επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε κάποια άλλα θέματα. Να είστε σίγουροι ότι η συνεργασία μας θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ε, αυτοκίνητο βιομηχανία. Εδώ από τη μία το ε, εμπόριο απειλείται με τιμωρητικούς δασμούς από την πλευρά των ΗΠΑ για παράδειγμα και εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε ε, ώστε να βρεθούν λύσεις που θα μας βγάλουν από, το, από αυτήν την κατάσταση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις αυτή τη στιγμή παρατηρούμε εξαιρετικά υψηλούς δασμούς για προϊόντα χαλιβουργίας. Όπως καταλαβαίνετε αυτό πλήττει και την βιομηχανία, αλλά οφείλουμε να δώσουμε την δέουσα προσοχή. Η Προεδρία μας έχει στόχο να προσπαθήσει να χτίσει γέφυρες έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, είναι προτεραιότητα της Προεδρίας μας, όμως ε, αυτό δεν είναι ευθύνη μόνο των ε, επιχειρήσεων. Χρειάζεται και χρόνος έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία να προσαρμοστούν ε, στις νέες απαιτήσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η ψηφιοποίηση αφορά πολλούς τομείς. Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα είναι ένα κεντρικός θεματικός άξονας. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται ολόνα και περισσότερο, από τη μία στην επεξεργασία δεδομένων, από την άλλη, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, αυτό θα είναι κάτι που θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Ε, είναι κάτι που αφορά την ίδια τη δομή της Ευρώπης. Γι' αυτό Πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο θα αφού θα προστατεύουμε τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, την στήριξη της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ερωτήσεις σας και ε, είμαι έτοιμη να απαντήσω σε επιπλέον ερωτήσεις και να είστε σίγουροι πώς θα φροντίσω η συνεργασία μας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις απαντήσεις σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Φάσμαν. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόλις έφυγε η κυρία Βαν γιατί ήθελα να της απαντήσω. Αλλά νομίζω πως ε, θα προσπαθήσω και χωρίς αυτό. Α, ναι, η κυρία Βαν Μπρέμτ έπρεπε να προετοιμαστεί για τον αγώνα μετά. Έξι ώρες μένουν, όμως εντάξει, ετοιμασίες είναι ετοιμασίες. Θα ήθελα όμω να απαντήσω στην ερώτησή τη ο κ. Υπουργό, ε, διότι είναι πολύ σημαντική. Η κυρία Βαν Πρέμπτ ε, αναφέρθηκε στην στρατηγική για ε, πολλού τομεί μέσα σε αυτού, είναι και έρευνα. Έχετε, έχει απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται στρατηγική, ερευνητική στρατηγική, χρειάζεται ενίσχυση των ε, τομέων όπου θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά χρειάζεται και προσοχή ε, στους τομείς που θα συνεισφέρουν στην κοινωνική ανάπτυξη. Ε, το Horizon Europe είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επιτευχθεί ιδιαίτερη, ιδιαίτερα καλή ισορροπία ανάμεσα στους πυλώνες, ανάμεσα στις ομάδες αυτές, τις επιμέρους ομάδες. αναφέρεται και σε θέματα ερευνητικά και Ίσως θυμάστε ότι αυτές οι, ομάδες, οι επιμέρους ομάδες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την ενέργεια, με την ασφάλεια, με μια ε, συνεκτική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα λοιπόν αυτά τα οποία προσπαθεί να απαντήσει και να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Επίσης ε, δίνεται έμφαση σε μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω με ε, προσοχή στην τόνωση της δημιουργικότητας. Είναι δύσκολο λοιπόν να, πούμε, να, να δούμε ποιες είναι οι στρατηγικά σημαντικές ε, στρατηγικά Το θέμα είναι η οπτική γωνία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στις πιο καινοτόμες προτάσεις και ιδέες και όπως σας είπα να σταθούμε στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Στον ορίζοντα Ευρώπη νομίζω πως υπάρχει μια καλή ισορροπία όλων αυτών. Η κυρία Βαν αναφέρθηκε και σε κάτι που ίσως δεν ανήκει οι απόλυτες αρμοδιότητες της Επιτροπής σας, όμως αναφέρθηκε στην ψηφιακή αλλαγή και στο ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να ε, αποφύγουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν θέματα απασχόλησης, υπάρχουν νέες προκλήσεις οι οποίες ε, απαιτούν μία επανακατάρτιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ψηφιακή αλλαγή. Και το δικό μου Υπουργείο, αλλά ε, νομίζω πως είναι γενικότερη η άποψη αυτή, θεωρεί πως αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα περισσότερο. Κύριε Κρασινοτέψκη, συγγνώμη που αν λέω λάθος το όνομά σας. Κάνατε επίσης δύο πολύ κέρια σημασίας ερωτήσεις. Η κυρία... Η Μαρή Κιουρί είχε κάνει πολύ σημαντικό έργο, χάραξε δρόμο πολύ δύσκολο. Εάν ζούσε η Μαρή Κιουρί, νομίζω πως ε, θα αναγνώριζε ότι χάρη σε εκείνη έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει πολλά βήματα έτσι ώστε να, α, να χτίσουμε βάσεις για το μέλλον. Επίσης η Mercury θα ήθελε αύξηση της χρηματοδότησης 1,5-2 δισεκατομμύρια παραπάνω. η έρευνα είναι η μηχανή της ε, οικονομίας μας και η συμπατριώτησά σας Εάν ζούσε το 2018 δεν θα χρειαζόταν ε, να ε, πετύχει στην δουλειά της ε, μέσω ενός γάμου διότι φυσικά η ισότητα έχει προχωρήσει. Τώρα, τα επιστημονικά project επιλέγονται με βάση την αξία τους και όχι με βάση το φύλλο. Έχουμε πάει λοιπόν μπροστά. Κύριε Γιάβορ, και εσείς έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για την Ευρατόμ και μάλιστα στη δική μας Προεδρία ε, μας είπατε ότι είναι δύσκολη για σας η ερώτηση, φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι για μας η απάντηση. Σίγουρα δεν έχει αλλάξει ε, η στάση μας. Η Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια είναι υπέρ μιας ε, ανανέωσης της συνθήκης Ευρατόμ. Διότι θέλουμε να κρατήσουμε τις επιτυχίες που αφορούν την προστασία από τη συνθήκη Ευρατών και να ε, διώξουμε τις ε, παροχημένες διατάξεις. Θέλουμε επίσης να ε, εκδημοκρατιστούν ορισμένες διαδικασίες. Αυτά είναι τα καλά. Όμως υπάρχουν και τα άσχημα. Ε, νομίζω πως δεν θα καταφέρουμε να ε, χειριστούμε το θέμα τη συνθήκης Ευρατών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αλλά θα λάβει τη σκητάλη η Ρουμανική Προεδρία και αυτό για ε, πολύ καλούς λόγους. Κυρία Κάπελ, κυρία Κάπελ δεν ξέρω αν είναι παρούσα. κυρία Κάπελ, θα ήθελα την ερώτηση σα να την απαντήσω ε, σε συνδυασμό με την ερώτηση του κυρίου Έλλερ. Γιατί και οι δύο ερωτήσει έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση. Το κατά πόσο τα 120 δισεκατομμύρια αρκούν ή όχι. Και θέλω να σα πω ότι αν ε, ξεπεράσουμε το ποσό των 100 δις, εγώ ακόμα καλύτερα για μένα. Προφανώς και δεν θα αντιδράσω. Ό,τι μου δώσουν θα το πάρω. Αλλά το θέμα του προπολογισμού είναι ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στι αρμοδιότητε του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εγώ θα υπερασπιστώ και την έρευνα και την καινοτομία. Ε, κυρίως και λιγότερο την ε, άμυνα, γιατί θεωρώ ότι με την έρευνα και την καινοτομία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Κυρία Κάπελ, εσείς ρωτήσατε επίσης ε, και νομίζω και η κυρία Βέρνικ και οι δύο το ποια είναι η διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και το Horizon Europe, ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ε, το, θα το δούμε, θα δούμε ποια ακριβώς είναι η διασύνδεση μεταξύ των δύο, αλλά εγώ τάσομαι ανεπιφύλεκτα υπέρ του να υπάρχει διασύνδεση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει προτάσεις. Πώς τη σκέφτεται αυτή τη διασύνδεση. Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν δώσει χρήματα για πάρα πολλέ γέφυρε, ε, για αυτοκινητόδρομους γιατί να μην δώσουν και για ερευνητικά και εδώ περιμένω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κύριε Ρουμπίχ, θέσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ερώτηση. Quantum Computing και HPC. Πώς ακριβώς συνδέονται αυτά τα δύο. Και οι δύο είναι τεχνολογίες του μέλλοντος. Αλλά η τεχνολογία HPC προφανώς και αφορά περίπλοκα τον υπολογισμό περίπλοκων μοντέλων προσωμείωσης, για να μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Η ε, φυσική σε σχέση με την HPC προσωμιώνει συνδέσεις μορίων έτσι ώστε για να δοκιμάζει υλικά. Και επειδή τα υλικά αποτελούνται από πολλές μοριακές συνθέσεις, χρειαζόμαστε τον υπολογισμό γιατί αυτό παίζει ρόλο στη φυσική. Τώρα, το computing, quantum computing είναι μια νέα μορφή τεχνολογίας και νομίζω και στις δύο περιπτώσεις η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει. Ειδικά στην τεχνολογία HPC, τι δεν μπορεί να κάνει το εθνικό κράτος, ξέρετε δεν μπορεί. Δεν μπορεί να επενδύσει σε τεχνολογίες κλίμακας, γιατί αν το καταφέρναμε αυτό ε, θα ήμασταν στη θέση 1000, 500 ή 1000 όσον αφορά τους μεγάλους υπολογιστές. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο υπολογισμού της Κίνας ή της Ιαπωνίας μόνοι μας. Αλλά αν τα συνδυάσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε και άσχημα. Και στο quantum computing και εκεί έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί ξέρετε στην αρχή δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς πόρους. Το quantum computing είμαι σίγουρος και επιμένω ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Ο κύριος Μπούζεκ με στραβοκοιτάει, ήδη με στραβοκοιτάει κοιτάει. Αλλά ξέρετε, επιτρέψτε μου να απαντήσω μια ερώτηση, να απαντήσω μια ερώτηση ακόμα. Ό,τι θέλετε, λέει ο πρόεδρος, απαντήστε ό,τι θέλετε. Γιατί αυτό που δεν θα απαντήσετε τώρα, θα το απαντήσετε εντό λίγο. Η δεύτερη συνάντησή μας, η συνεδρίασή μα συνεχίζεται και πάλι με εσά. Εγώ όμως θέλω να απαντήσω στην κυρία Μόντε σχετικά με το κενό που υπάρχει στην εφαρμογή ερευνητικών συμπερασμάτων, συμπεράσματα που έχουν σχέση με την κοινωνία. Και έχετε απόλυτα δίκιο, πράγματι εδώ υπάρχει ένα κενό, είμαστε πιο πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό και με τις διοικητικές διαδικασίες. Δηλαδή πότε μπορεί κανείς, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιο κόστος να στηρίξει να ιδρύσει μια εταιρεία. Και κάποιος που ιδρύει μια εταιρεία, τι είδου ευθύνε αναλαμβάνει. Μήπως ε, θα ήταν καλύτερα ο άνθρωπος αυτός ε, να είναι υπάλληλο μια εταιρεία και όχι ανεξάρτητος και αυτοδημιούργητος επαγγελματίας. Εκεί στις ΗΠΑ Πολιτείες τα πράγματα είναι πολύ, απλά, πολύ πιο απλά. Όμως το πρόγραμμα Horizon το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα και ο πυλώνας 3 κάνει ακριβώς αυτό. Pathfinding λέγεται. Δηλαδή αναζητούνται ενδιαφέρουν σε ε, τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει μια τομή, μια πραγματική τομή. Και επίση αναζητούνται και για χρηματοδοτικές δυνατότητες για spin-offs, spin-offs που θα διονγκωθούν. Σε αυτόν λοιπόν τον τρίτο πυλώνα που αφορά την καινοτομία πρέπει να συζητήσουμε με την Κομισιόν γιατί και εγώ ίδιος δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Δηλαδή πώς μπορώ να βρω αυτές τις ε, νέες τεχνολογίες. Μπας περιπτώσει έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο και μπορούμε να συζητήσουμε αυτό που είναι το βασικό είναι να υπάρχει το θέμα στο θεματολόγιο. Το, το θεματολόγιο να υπάρχει research and impact οι προεκτάσεις, όλα αυτά τα θετικά που προκύπτουν από την έρευνα. Και να απαντήσω και άλλη μια ερώτηση για να μην την απαντήσω αργότερα. Απευθύνομαι στον κύριο Σορίνο, Σορίνιο, ο οποίος ρώτησε είπε το εξή. Σήμερα μιλήσατε, αν κατάλαβα καλά, για την ενεργειακή απόδοση και πώ να αντιμετωπίζει η έρευνα. Θέλω να σα πω ότι η ενέργεια είναι ένα στρατηγικό ερώτημα. Κλάστερ 3, πυλώνο 2, 15 δι θα δαπανηθούν για την ενεργειακή έρευνα. Αυτό είναι μια ανακοίνωση. Και βεβαίω μπορεί κανείς να περιμένει ε, οι εθνικοί θεσμοί και τα κράτη να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση, να προσαρμοστούν. Και αυτό σημαίνει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα 15 δις θα πολλαπλασιαστούν τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά μας Ινστιτούτα θα προσαρμοστούν και θα ακολουθήσουν αυτό που αποκαλούμε στην έρευνα alignment. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς. Ήταν ε, πολύ καλή ευκαιρία για μας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε ανοιχτά τόσο σημαντικά θέματα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία γιατί εξαρτώνται πάρα πολλά από την Προεδρία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την ε, ανοιχτότητά σας εδώ και κάθε επιτυχία σας εύχομαι.

Κυρίες και κύριοι, κάποια θέματα. Αναφέρθηκαν ε, κάποιες ερωτήσεις για θέματα ενέργειας. Όμως και πάλι θα έχουμε τώρα τον Υπουργό Χάιν Φάσμαν, ο οποίος αντικαθιστά την Ελίζαμπεθ Κέστιγκερ. Ομοσπονδιακή Υπουργό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Τουρισμού της Αυστρίας και γενικώ και για την ενέργεια. Ορισμένε από τι ερωτήσει απαντήθηκαν, επομένως δεν είναι απαραίτητο να τι ξαναθέσουμε επιτάπητο, αλλά και εγώ έχω μια ερώτηση για την ενέργεια. Βέβαια δεν την έθεσα πριν. Όμως, κύριε Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας δώσουμε το λόγο για να ξεκινήσετε. Από ό,τι καταλαβαίνω, κατά τη διάρκεια της ε, Αυστρικής Προεδρίας, οι δικές σας αρμοδιότητες, αλλά και της ε, κυρίας Κέστικερ, θα συμπεριλαμβάνουν το πακέτο καθαρής ενέργειας, το ενεργειακό τμήμα του προγράμματος Συνδέοντας ε, την Ευρώπη, του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη και επενδυτικά project σε ενεργειακές υποδομές. Πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν αυτά για την Επιτροπή μας. Καθώς είμαστε καθολικά αρμόδιοι για τα ενεργειακά ζητήματα ως Επιτροπή. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Αξιότιμε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να μπορώ εδώ να σας ε, απευθύνω το λόγο. Ε, αντικαθιστώ την κυρία Κιώστιγκερ η οποία από την Κυριακή είναι μητέρα, έγινε μαμά του Λόρεντς Ιωάννης του Μπέμπι. Και επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τους ε, χαιρετισμούς της. Um, ich möchte mich auch bedanken bei θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Πέτκοβα ε, από τη Βουλγαρία και την Υπουργό από την Εστονία. Να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους αδέλφους από τη Βουλγαρία και την Εστονία, οι οποίοι ε, στα πλαίσια της ε, Τρόικα, Προεδρία Τρόικα, συνέβαλαν και αυτοί πάρα πολύ στις εργασίες μας. Νομίζω ότι στους τελευταίους μήνες πετύχαμε μεγάλη πρόοδο και κατά κάποιον τρόπο εναπόκειται τώρα στην Αυστρία να συνεχίσει την πρόοδο αυτή. Με την κυρία Κιώστιγκερ ε, ω Υπουργό Ενέργεια, γιατί εντάξει, σύντομα θα αναλάβει και πάλι το έργο της Κατά τους επόμενους έξι μήνες θα έχουμε ε, κινητήρια δύναμη για, την, ε, για το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ενέργειας. Και θέλουμε να είμαστε τίμοι διαμεσολαβητές και τα δικά μας τα συμφέροντα να τα βάλουμε σε τρίτη θέση. Ο στόχος της περαιτέρω ανάπτυξης ε, είναι να έχουμε μια ισχυρή ενεργειακή ένωση η οποία θα είναι προϋπόθεση για να έχουμε ένα ανταγωνιστικό βιώσιμο σύστημα ενέργειας. Επίσης αυτό που θέλουμε είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ενταχθούν καλύτερα στο όλο πρόγραμμα. Είμαστε επίσης ε, αισιόδοξοι ότι θα έχουμε επικοδομητική συνεργασία με όλους τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε επίσης ότι η μέχρι τώρα άποψη που, που κρατεί αυτή, η ολιστική άποψη για την ενέργεια και την κλιματική πολιτική, αυτή η άποψη είναι σημαντική. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ε, θα έχουμε τρία βασικά θέματα. Ε, το καθαρό πακέτο, δηλαδή θέλουμε να επιδιώξουμε το να ολοκληρωθούν ε, όλες οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν αυτό το, το πακέτο της καθαρής ενέργειας. Και θέλουμε βέβαια να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα. Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διάλογοι για τους ε, για το καθαρό ενεργειακό πακέτο και οι τρεις αυτοί τριμερείς διάλογοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Έχουμε τον κανονισμό για τη διαχείριση, για την ενεργειακή απόδοση και έχουμε και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που επίσης επιθυμούμε είναι να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές ε, για τα θέματα αυτά, Τουρμές, Πόχε και τον κύριο Χωσέ Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστούμε και τους τρεις, γιατί και οι τρεις ε, παρουσίασαν ε, πολύ καλή εργασία, από κοινού βέβαια με την Βουλγαρική Προεδρία. Και επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου να τράξω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά που επιτύχατε και κυρίως και για την προθυμία που επιδείξατε για την επίτευξη συμβιβασμών. Με την ολοκλήρωση και θέσπιση αυτών των νομοθετικών πράξεων επιτεύχθηκε θέμενη αξία στην Ευρώπη. Οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ σημαντικοί και γενικά εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη για την ε, συνάντηση COP24 στο Κατόβιτσο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη. Τα θέματα τα οποία ε, παραμένουν είναι κυρίως ο σχεδιασμός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ε, θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια εφοδιασμού και με τις ρυθμιστικές αρχές. Όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα που προβλέπονται στη Συμφωνία των Παρισίων θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον ανασχεδιασμό της κοινή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως τμήμα της καθαρής ενέργειας ε, για το ενεργειακό πακέτο, ο κανονισμός ε, της κοινή αγοράς ε, για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η σχετική οδηγία, είναι καθοριστική σημασίας για την εξέλιξη της, ε, ηλεκτρικής, ε, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κυρίως όσον αφορά τον κανονισμό, εκεί η Αυστρία θα προσπαθήσει να βρει εφικτές λύσεις που θα ωφελήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά και το να παραμείνει η Ευρώπη έδρα των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν βέβαια επίμαχα θέματα, έτσι μου έχουν πει, ε, προς τα δεξιά στρέφω το βλέμμα και έχω κάθε λόγο που το κάνω αυτό. Υπάρχει το θέμα των μηχανισμών ε, δυναμικότητας και αυτό είναι ένα επίμαχο θέμα. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν είναι να καταλήξουμε σε ικανοποιητικούς κανονισμούς οι οποίοι θα είναι συμβατοί και με τις ρυθμίσεις για την κλιματική αλλαγή. Η ε, δημιουργία ίσων προϋποθέσεων για όλους που συμμετέχουν στην κοινή αγορά. Αυτό επίση είναι ένα στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε με τον κανονισμό, με τη θέσπιση του κανονισμού. Πέρα από αυτό, αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να ισχύσουμε και ε, τα δικαιώματα του καταναλωτή. Έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων προς όφελος των πολιτών. Στην ε, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ε, να μπορούν να συμμετέχουν διάφοροι φορείς και πιστεύουμε αυτό είναι ένας ουσιαστικός στόχος και ένα καθοριστικό σημείο για να επιτευχθεί ενεργειακή αλλαγή, μια καμπή στην ενέργεια. Και, και τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως ε, προβλέπεται και αντιμετώπιση κινδύνων που έχουν σχέση με την ενέργεια. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση και για τον κανονισμό και για την οδηγία που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί στην περίπτωση που έχουμε εύρυθμα λειτουργούσες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, εκεί το μόνο που μπορεί να υπάρξει είναι ένας κίνδυνος εφοδιασμού. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και γι' αυτό οφείλουμε να μεριμνήσουμε με προληπτικά μέτρα. Και τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί σήμερα η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ε, πλέον είναι διασυνοριακή. Έχει τέτοιου είδους χαρακτήρα και οι, εφοδια... οι κρίσεις εφοδιασμού σε ένα κράτος μπορούν κάλλιστα να έχουν επιπτώσεις και σε άλλα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ένα πανευρωπαϊκό, ένα ενωσιακό εργαλείο έτσι ώστε να αποφεύγονται κρίσεις εφοδιασμού. Η Αυστρία σε αυτό το θέμα θα προσπαθήσει ε, να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα διασφαλίζει ή θα αυξάνει περισσότερο την ασφάλεια. Ένα άλλο θέμα που θα, το θα απελευθούμε είναι ο οργανισμός εκείνος που αφορά στη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών, ACER και αυτός ε, ο φορέας έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία ε, στο πλαίσιο του ε, πακέτου καθαρής ενέργειας για όλους. Προβλέπεται η προσαρμογή των φορέων στην πραγματικότητα και κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες. Η Αυστριακή Προεδρία έχει πολλές φιλοδοξίες. Θέλουμε να επιτύχουμε μια ισόρροπη λύση. Μια λύση που θα επιτρέπει όμως να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη, να λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους. Μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα αλλά και η διασφάλιση των πόρων και της επικουρικότητας. Το πρόγραμμά μας ή το πρόγραμμά σας αν θέλετε είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πολύ συμπυκνωμένο. 17 και 18 Σεπτεμβρίου έχουμε άτυπη, άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λίντς και εκεί έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε για να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο. Ε, κυρίως ε, όσον αφορά αυτά τα εναπομέναντα νομοθετικά θέματα. Ένα άλλο θέμα που αφορά στην Προεδρία μας είναι η οδηγία περί εσωτερικής αγοράς αερίου. Υπό την Βουλγαρική Προεδρία έγιναν πολλές συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Υπήρξαν πολλές και διαφορετικές θέσεις και υπήρξαν επίσης και κάποια ε, νομικής και τεχνικής φύσεως θέματα που εφήγησαν. Γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό έχει μεγάλη πολιτική σημασία για αρκετά κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία έχει ε, επιβραδυνθεί η Κορεπέρ, επειδή υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα, ανέπεμψε το θέμα σε τεχνικό επίπεδο. Εμείς θα συνεχίσουμε την εξέταση του θέματος. Γνωρίζουμε ότι από πλευράς Κοινοβουλίου υπάρχει κάποια προθυμία έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι δύο οργανικές διαπραγματεύσεις. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα για μας είναι οι καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες. καινοτομικές Προφανώ προφανώς και είναι κλειδί ε, για να επιτύχουμε την ενεργειακή ένωση. Και στο άτυπο ε, Συμβούλιο Υπουργών 17 ε, και 18 Σεπτεμβρίου που σας ανέφερα προηγουμένως εκεί θα εξεταστούν καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες. Το σύνθημά μας είναι Charge for Change που νομίζω έτσι είναι ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά πολύ ενδιαφέρον και υπονοεί να αποδοθεί σημασία στο υδρογόνο, στις ε, τεχνολογίες δέσμευσης ε, και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ενεργειακή καμπή. 20 και 21 Νοεμβρίου θα έχουμε την 11η συνεδρίαση η οποία και αυτή θα ασχοληθεί με θέματα εναλλακτικών τεχνολογιών η συνδύση του Άσερ. Και αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι να έχουμε ανθεκτικά κτίρια ενεργειακά ενδιαφέροντα κτίρια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί ξέρετε μπορεί κανείς να εξοικονομήσει όση ενέργεια θέλει. Αλλά αν υπάρχει τέτοια πολεοδομία η οποία οδηγεί σε χρήση μεγαλύτερων όγκων ενέργειας, τι να την κάνετε την εξοικονόμηση. Σημαντικό για μας είναι η ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία, αλλά και κοινά προγράμματα που αποδίδουν τη θέμενη αξία, έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 και επίσης και να υπάρχουν οι δυνατότητες χρηματοδότησης της νέας ενεργειακής πλατφόρμας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις 27 Απριλίου έλαβε χώρα ένα, μια ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου στη Βιέννη. Και εκεί τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο, γιατί το Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Κλώτο Τουρμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού ΕΦΣΙ, ο κύριος Μόλτερ, επέδειξαν όλοι αυτοί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτό τον ενθουσιασμό έτσι ώστε και με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία να μπορέσουμε να προσελκύσουμε χρηματοδότηση για προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα άλλο τρίτο θέμα, International Energy Hub Austria. Αυτό τι είναι. Είναι μια προσπάθειά μας για να ενισχύσουμε το διάλογο και πέρα από τα εθνικά όρια. Πιστεύουμε ότι η Βιέννη η Αυστρία, αν θέλετε, είναι καταδικασμένες, αν μου επιτρέπετε να πω, να πράξουν κάτι τέτοιο. Γιατί, Γιατί στη Βιέννη έχουμε πολλούς διεθνείς οργανισμούς που έχουν σχέση με την έργεια. Την UNIDO, την ε, Sustainable Energy for All, την ε, Ενεργειακή Ένωση για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ε, αυτό λοιπόν το ότι είναι όλοι αυτοί οι διεθνεί οργανισμοί στη Βιέννη το βρίσκουμε ατού. Και στι 15 ε, Νοεμβρίου θα συναντηθούν οι γενικοί διευθυντέ αλλά και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Υπουργείων ε, θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών για να συζητήσουν για την ενεργειακή ασφάλεια την εποχή της κατάργησης χρήσης του άνθρακα και χρήσης περισσότερων καινοτόμων μορφών ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, εκτός αυτού η Αυστριακή Προεδρία ε, σε όλα τα επίπεδα θα επιδιώξει την πιο ουσιαστική συνεργασία με τα Βαλκάνια βρισκόμεθα αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Θα τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Και χαιρόμεθα, αυτό δεν είναι μια κοινότοπη φιλοφρόνηση, χαιρόμεθα πραγματικά που θα μπορέσουμε κατά τους επόμενους έξι μήνες να συνεργαστούμε με πολλού η φιλοδοξία μας είναι να επιτύχουμε πρόοδο έτσι ώστε να επιδιώξουμε μια αηφόρο αγορά ενέργειας που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές και θέλουμε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε, που μου δώσετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις προτεραιότητές σας και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μου υποβάλλετε ερωτήσεις. Και θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, με την ευχέρεια το οποίο θα είχε να απαντήσει η καθήλυνα αρμόδια υπουργό, η κυρία Κιώστιγκερ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να πω πολύ ανοιχτά, γιατί είμαστε πολύ ανοιχτοί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η ομιλία σα ε, ήταν ε, ιδιαίτερα μακροσκελής, δύο φορέ πιο μακροσκελής από ό,τι περιμένουμε. Αλλά είναι εντάξει, γιατί πρόκειται για μια παρουσίαση εκ μέρου ε, τη συναδέλφου σα, τη κυρία Κέστιγκερ, που δεν είναι εδώ παρούσα. Έτσι λοιπόν, ε, κατανοούμε ότι μπορούν να είναι πολύ σύντομες οι απαντήσεις σας. Το σημαντικό για μας είναι να θέσουμε τις ερωτήσεις μας, τις παρατηρήσεις μας ε, και τις αμφιβολίες μας ε, για να τις διαβιβάσετε στη συνάδελφο στην Αυστριακή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι οι απαντήσεις σας μπορεί να μην είναι αντίστοιχε στον προσδοκιό μας. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι δεν είστε αρμόδιος ε, για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ήταν ε, πολύ πληρή η παρουσίαση, εξαιρετικά. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Θέλω να ζητήσω και από τους συνάδελφου να είναι όσο δυνατόν πιο σύντομοι, γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Στις 6 και μισή ακριβώς θα θέλαμε να τελειώσουμε. Και θα έχουμε ακόμη πέντε σημεία στην ημερησία διάταξη και το ένα είναι το πρόγραμμα πλαίσιο, πολύ σημαντικό. Δύο μέρη του προγράμματος πλαισίου. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα και δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε ένα λεπτό παραπάνω, όπως ξέρετε. Γιατί δεν θα έχουμε διερμηνία μετά τις 6.30. Λοιπόν, περνάμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, όσο το δυνατόν πιο σύντομη να είστε. Από το ΕΛΚΟ, κύριος Κάρνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχω ερώτηση, περισσότερο σχόλιο. Εγώ είμαι εισηγητής ε, για την οδηγία και τον κανονισμό περισχεδιασμού της ε, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας ε, θα μπορέσετε να πετύχετε ένα συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκατε στο μηχανισμό δυναμικότητας, είναι ένα από τα επίμαχα ζητήματα, αλλά υπάρχουν αρκετά και στον κανονισμό και στην οδηγία, το πώς θα αντιμετωπίσουμε και την ενεργειακή ανέχεια. Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε αυτά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί να βρούμε ένα κοινό τόπο αν ε, το Κοινοβούλιο έχει μία ενοποιημένη άποψη για το πώς θα είναι το κείμενο, δηλαδή μια ισχυρή εντολή, φαίνεται ότι το Συμβούλιο είναι αρκετά διαιρεμένο. Υπάρχει διχογνωμία στο Συμβούλιο. Και αναφερθήκατε και στην οδηγία για το αέριο. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε κάποια διέξοδο από το διέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε στο Συμβούλιο μέχρι τώρα θα θετήσετε μια νέα προσέγγιση. Εμείς ε, από τη σκοπιά μας, από την πλευρά μας, εργαζόμαστε πολύ σκληρά. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Μπούζε, κάθεται δίπλα σας. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει ε, μία πρόοδος. Έχουμε ευρωπαϊκό δίκαιο που διέπει τις ευρωπαϊκές επιδομές. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το δίκαιο θα έπρεπε να ισχύει σε όλε τι υποδομέ. Πώ ε, λοιπόν θα βγούμε αυτό το διέξοδο και θα σημειωθεί πρόοδο. Σα ευχαριστώ πολύ ο κύριος ε, Πλανκολόπες για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εργαζόμαστε πάνω από ένα μισή χρόνο στο Ινέδεσμο Μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια στο Κοινοβούλιο, το μεγαλύτερο πακέτο μέτρων για την ενεργειακή μετάβαση τα επόμενα έτη. Κατά τη διάρκεια τη Βουλγαρική Προεδρία, ε, συμφωνήσαμε σε τρία μεγάλα καρτοφυλάκια αποδοτικότητα, ανανεώσιμε και διακυβέρνηση. Και τώρα εσεί ε, θα πρέπει να ε, έχετε αντιμετωπίσετε την μεταρρύθμιση του σχεδιασμού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, χρειαζόμαστε για τους συμβιβασμού ε, κάποια νομικά πλαίσια που να τα υλοποιήσουν και θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τι ενέργειε που προέρχονται από ρηκτά κόψιμα με έσχημε πηγέ ενέργεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε στην τύχη του ε, τι περιοχέ ε, των οποίων ε, η οικονομία σχετίζεται με τέτοιε δραστηριότητε. Το αντίθετο, θα πρέπει να του προσφέρουμε εξόδου, διεξόδου για ένα νέο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποιε είναι οι προτεραιότητε τη δική σα Προεδρία ω προ τον κανονισμό και την οδηγία για το σχεδιασμό τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερον, πώ θα προσεγγίσετε την μείωση των εκπομπών άνθρακα μέσω μια δίκαιη μετάβαση που θα λαμβάνει υπόψη και την ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Και ε, γνωρίζω ότι η υπουργό ξέρει πάρα πολύ ε, καλά αυτό το φάκελο και μάλιστα είχε καταθέσει και τροπολογίε ω Ευρωβουλευτή. επομένω νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλά χέρια. Ευχαριστώ. Από το ECR ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να επανέλθω στην ερώτηση. Έχουμε ήδη μιλήσει για το θέμα αυτό. Όμως, η Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί με το θέμα της οδηγίας της αναθεώρησης του αερίου στις επόμενες συνεδρίες της Κορεπέρνα ή όχι. Και το γεγονός ότι μία από αυτές τις μεγάλες αυστριακές επιχειρήσεις συμμετέχει στο Nord Stream 2 δεν θα σας θέσει εμπόδια στο να το πράξετε αυτό. Εγώ ελπίζω να μιλήσουμε για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν μία σειρά δύσκολων σημείων ε, και που είναι ακόμα εκκρεμή. Παραδείγματο χάρη η διαφορετική μεταχείριση του μηχανισμού της αγοράς ε, και των στρατηγικών αποθεμάτων. Όμως είναι επίσης πολύ σημαντικό το θέμα των ε, περιοχών των τιμών και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι συζητείτε πολύ αυτό το θέμα στην Αυστρία και θα ήθελα να μου πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Εμείς ε, θα θέλαμε να παρέμβει η Προεδρία σε αυτό το θέμα, κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για τις παρατηρήσεις του. Τώρα όλοι θα είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Όχι μόνο με τους φακέλους που αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους για το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Από όσα κατάλαβα από την εισαγωγή σας, είπατε ότι οι σημερινές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκφύσιως διασυνοριακές. Αυτό θα ήθελα κάπως να το αμφισβητήσω. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι μόνο το ίμιση της Ευρωπαϊκής Διασυνορικής Δυναμικότητας ε, χρησιμοποιήθηκε πέρσι. Έτσι, λοιπόν, η πρόκληση δεν είναι ότι είναι εκφύσεως διασυνοριακή, αλλά ότι δεν έχουμε επαρκείς διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ή ενέργειας αυτής καθ' Και νομίζω ότι είναι απολύτως ε, κρίσιμο για την Αυστριακή Προεδρία να έχει μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αγορά όπου θα τονίσετε τη σημασία του να πετύχουμε διασυνοριακές ροές στην ηλεκτρική ενέργεια γιατί δεν έχουμε εσωτερική αγορά ενέργειας σήμερα και φυσικά αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις, είναι υψηλότερες οι τιμές από ό,τι θα έπρεπε δεν ε, πετυχαίνουμε τους στόχους μας, ε, τους κλιματικούς, ούτε σεβόμαστε τη Συμφωνία των Παρισίων. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δίκτυά μας αν είχαμε περισσότερες διασυνοριακές ροές. Και έχουμε και μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα στις ζητήσεις με το Συμβούλιο ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι πολύ απλά. Αν εσείς θα έχετε μία προσέγγιση που να βασίζεται στην αγορά για το θέμα αυτό, θα δώσετε περαιτέρω έμφαση στη σημασία των διασυριακών ανταλλαγών ενεργειακών γιατί αυτό θα μπορούσε να έχει μια μεγάλη σημασία και να κάνει τη διαφορά για όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ για τους Πρασίνους, ο κύριος Κιάβο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω το θέμα του μηχανισμού δυναμικότητας και του σχεδιασμού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα. Με ενδιαφέρει κυρίως η θέση της Αυστρίας. Γιατί το Κοινοβουλίο και η Κομισιόν κατά κάποιο τρόπο έχουν δεσμευτεί στο να εφαρμόσουν τους μηχανισμούς δυναμικότητας ε, με έναν ε, πιο περιορισμένο τρόπο για να ε, ενθαρρύνουν το διασυνορική φύση του μηχανισμού δυναμικότητας και επίσης να υπάρχουν και όρια εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στο μηχανισμό δυναμικότητας. Όλα αυτά αντιφυσβητούνται όμως από κάποια κράτη-μέλη. Συμφωνώ λοιπόν με τους συναδέλφους ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια συνένεση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Επομένως, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η θέση της Αυστρίας για τα θέματα αυτά. Τη διασυνοριακή φύση του μηχανισμού δυναμικότητας, ε, τα όρια των εκπομπών του άνθρακα κτλ. Επίσης, για την οδηγία του αερίου. Αυτό σχετίζεται με το θέμα του αγωγού Nord Stream 2. Και εκεί θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση του επόμενου μήνε. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Από την ΚΟΕ, ο κύριο Ηλικιώτης. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, εγώ θα ξεκινήσω από ένα θέμα που ε, δεν σχολιάστηκε μέχρι τώρα. Για όλους μας θα έπρεπε η ενέργεια να αποτελεί ένα βασικό δημόσιο αγαθό, να υπάρχει δηλαδή καθολική πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Το πρώτο θέμα που ήθελα να θέσω ως ερώτημα είναι τι προτίθεται να κάνει η Αυστριακή Προεδρία για να στηρίξει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για προστασία και ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού τη αγορά ενεργεία, για διασφάλιση δηλαδή τη πρόσβαση σε ολοκληρωμένη ενημέρωση, για συμβόλαια στη βάση των αναγκών των καταναλωτών, για διαφάνεια, για στήριξη ιδιαίτερα των καταναλωτών από ευάλωτε ομάδε. Το δεύτερο αναφέρεται στο πρόγραμμα τη Αυστριακή Προεδρία ο στόχο για ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία και στον τομέα τη ενέργεια. Πέραν όμω τη ανταγωνιστικότητα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εδώ στην Επιτροπή το συζητήσαμε πολλέ φορέ. Είναι το πρόβλημα τη ενεργειακή στόχια. Εκατομμύρια συμπολίτε μα σήμερα στην Ευρώπη συγκαταλέγονται στην ομάδα τη ενεργειακή στόχια. Τι είναι αυτό που θα προτείνει ή θα συζητήσει η Αυστριακή Προεδρία ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να στηριχτούν οι ευάλωτε ομάδε και εκείνε η μερίδα του πληθυσμού που κατάσταται στην ενεργειακή φτώχεια ε, και θα μπορούσε η Αυστριακή Προεδρία να προωθήσει ένα ε, κοινό ορισμό τη ενεργειακή φτώχεια στη βάση ενό συνόλου κριτηρίων για μέτρηση τη ενεργειακή παινία. Μια κριτική που ασκούμε μέχρι σήμερα ότι ούτε από το Συμβούλιο ούτε από την Επιτροπή, ενώ γίνεται αναφορά στην ενεργειακή φτώχεια, δεν υπάρχουν μπροστά μα συγκεκριμένε προτάσει. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω είναι κατά πόσο η Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί με τα θέματα των εχώριων πηγών της Ένωσης των ενεργειακών πηγών. Ε, γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση και σήμερα υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και αναφέρομαι στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κυπριακή Ναός και στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά πόσο υπάρχουν κάποιες σκέψεις πώς θα προωθήσει το θέμα ώστε να αξιοποιηθούν αυτές οι νέες πηγές ενέργειας που ανακαλύφθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, e Η κυρία Κάπελ από ENF. Ο συνήθως. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Φάσμαν, τα τρία σημαντικότερα ε, θέματα του τομέα της ενέργειας ήδη αναφέρθηκαν το δεσμέτρων για την καθαρή ενέργεια, το διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη που θα συμπεριληφθεί στο επόμενο πού και οι ενεργειακές υποδομές και επενδύσεις. Στην Επιτροπή Ήδη έχουμε ψηφίσει τρία, τρεις εκθέσεις για ε, το πρώτο θέμα, την ενεργειακή απόδοση, η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ήδη αναβαρθήκατε και στην εσωτερική αγορά ενέργειας, οδηγία και κανονισμός με έμφαση στην, στους μηχανισμούς ε, δυνατοτήτων και Acer και αγορά ενέργειας. Είναι τρία πολύ σημαντικά θέματα για την εσωτερική ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η εσωτερική αγορά αερίου είναι κάτι που ε, μας απασχολεί. Είναι πολύ σημαντικό. Η, το Connecting Europe θα πρέπει να θα πρέπει να λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μόνο και μόνο για την ανάπτυξη υποδομών, ενέργειας, αλλά και θα πρέπει να ε, δοθεί επαρκής ε, χρηματοδότηση στις ε, διασυνδέσεις της ενεργειακής. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι, ε, θεωρείτε πως είναι ρεαλιστικά τα σχέδια. Ξέρετε πως ε, μέχρι το 2020 πρέπει να αυξηθεί κατά 10% και από το 2020 έως το 2030 κατά 20% η συνδεσιμότητα. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε συνοπτικά τα νέα έργα, τα νέα project και, ε, που αποσκοπούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια παράκληση περισσότερο παρά ερώτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το, την υπηρεσία ΣΤΟΑ και ασχολείται με θέματα ενέργειας και τεχνολογίας διεξάγει μελέτες, εκτέσεις, εκτιμήσεις. Υπάρχει αρκετή γνώση που έχουν συλλέξει, όμως ε, δεν ε, αναφέρεται κάποια στρατηγική επικοινωνίας. Ακούσαμε για την τεχνητή μοημοσύνη, για την ε, χρήση των, του μεγάλου όγκου δεδομένων, big data. Όμως υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία σε αυτό. Επίσης, ο Μπέρεκ, ο οργανισμός ε, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και ο Acer, ο Οργανισμός για την Αγορά Ενέργειας, καθώς και ο ENISA για την προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια ε, κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των ε, αυτών οργανισμών, μεταξύ των ε, διαφόρων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω σε εσά να αναλάβετε πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Ήταν όλες πολύ σημαντικές. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Ναι, ναι, ε, σήκωσα το χέρι μου στην αρχή, αλλά μάλλον ήταν πολύ μικρό και δεν με είδατε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φρόιντ έχει το λόγο, λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, και Φασμαν, δεν θέλω να σας καταστήσω υπεύθυνο, όμως ε, στην Αυστρία έχουμε πρόβλημα αξιοπιστίας σε ό,τι φορά τους ε, στόχους για το κλίμα. Αλλά και σίγουρα ε, το θέμα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην Αυστρία και έχουμε δυστυχώς ε, αποτύχει σε όλους τους σχετικούς ε, στόχους. Γι' αυτό λοιπόν όταν ακούω ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, στοχεύουμε σε αυτό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω λόγω του προηγούμενου. σήμερα όμως ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά θα με ενδιαφέρει να μάθω περισσότερα για τον ΙΤΕΡ, τον ε, πειραματικό ε, αντιδραστήρα στην Γαλλία. Τι γνώμη έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ για, όλη, για την ερώτησή σας. Και να προσθέσω κάτι. Ε, κάτι ως συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης. Είπατε εκ μέρους της κυρίας Κόστινγκερ ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι καθοριστική σημασία για την αγορά ενέργειας και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό της αγοράς ε, ηλεκτρικής ενέργειας, ε, την ε, σχετική οδηγία και τον κανονισμό. Μας λείπουν οι ορισμοί, ένας πολύ βασικός ορισμός των διασυνδέσεων, interconnectors, στην οδηγία. Πρέπει να τελειώνουμε το συντομότερο, όπως είπατε κι εσείς. Στην αναθεώρηση της οδηγίας για το αέριο υπάρχει ένας ε, παρεμφερής ορισμός της γράμμης διασύνδεσης, του interconnector. Παρόμοιος. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Πώς σκοπεύετε να εναρμονίσετε τη δουλειά σε αυτές τις δύο σχετικές οδηγίες. Γιατί. Αν διαφωνείτε με τον ορισμό των ε, γραμμών ε, διασύνδεσης και αν έχετε τόσες πολλές αμφιβολίες ε, εκεί στο Συμβούλιο, θα είναι σχεδόν αδύνατο να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για την νομοθεσία σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς θέλουμε να σας παροτρύνουμε να ξεκινήσετε μια σοβαρή συζήτηση για την αναθεώρηση της οδηγίας για το αέριο, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι νωρίτερα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, με χαρά λοιπόν να ακούσουμε τις, ελπίζω σύντομες απαντήσεις σας, αλλά ίσως πιο σημαντικό, θα θέλαμε να μεταφέρετε στην ε, συνάδελφό σας, την κυρία Κόστινγκερ, την Υπουργό Τουρισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ε, αλλά και Ενέργειας, ε, τις ερωτήσεις μας. Ξέρουμε πως θα συνεργαστείτε το επόμενο εξάμεινο για πολύ σημαντικά θέματα, όπως η αγορά ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι θα μεταφέρω τις ερωτήσεις στην ε, συναδελφό μου και επίσης ε, θα τις μεταφέρω τις εντυπώσεις που αποκόμισα από τη συζήτηση σήμερα. Κύριε Κρασινοντέμψκη, να αρχίσω με τη δική σας ερώτηση πρώτα σχετικά με την, εσωτερική, με την οδηγία για την εσωτερική αγορά αερίου. Στην Κορεπέρ φάνηκε ότι δεν υπάρχει συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν ως απάντηση μπορώ να πω ότι πρέπει να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις τις σχετικές, στο σχετικό πλαίσιο και να δούμε πώς θα επιτευχθεί αυτή η συνένεση. Κύριε Κάριντς, νομίζω είστε υπερβολικά αισιόδοξο για τη διαπραγματευτική ικανότητα της ε, Αυστηρικής Προεδρίας. Ελπίζω να μπορέσουμε να ανταπεκριθούμε στις προσδοκίες σας. Υπάρχει πολυμορφία στη μεταφορά φυσικού αερίου από διάφορες χώρες. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Όμως σίγουρα αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με την εναρμόνιση των διαφόρων έργων υποδομής. Κύριε Πέτερσεν, μιλήσατε για διασυνοριακές ανταλλαγές ε, ε, σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, πως δεν χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο έπακρο, στον κανονισμό για την ιστορική αγορά ενέργειας, στα πλαίσια του τριμερού σε διαλόγου σίγουρα χρειάζεται φιλοδοξία, διότι θέλουμε να είμαστε βασισμένοι στην αγορά. Πιστεύουμε στην αγορά, μεν, αλλά πρέπει να προσέξουμε και τον ε, ενεργειακό εφοδιασμό. Και χρειάζεται επομένως ε, κάποια αρρύθμιση στην αγορά. Κύριε Κάριντς και κύριε Γιάβορ, αναφέρατε και οι δύο τις ε, δυνατότητες, τους μηχανισμούς τους οικονομικούς που θα εγγυηθούν αυτήν την ισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει λοιπόν αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ε, ενεργειακή ασφάλεια. Ασφάλεια του εφοδιασμού, συγγνώμη. Σίγουρα πρέπει να γίνονται σεβαστά κάποια όρια και πρέπει να θεσπιστούν όρια για το πόσο διοξίδιο του άνθρακα επιτρέπεται να ε, εκλεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Αυτό θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί, διότι όπως ξέρετε οτιδήποτε έχει να κάνει με νομοθεσία και θέσπιση ορίων είναι κάτι πολύ δύσκολο. Κύριε Σιλικιώτη, αναφερθήκατε στην ενεργειακή ένδυα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ε, επίσης πολιτικά επίκαιρο. Ήθελα όμως να πω ότι τα εθνικά συστήματα στήριξης είναι τα πρώτα που θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για το θέμα αυτό. Ε, πρώτα δηλαδή το εθνικό επίπεδο πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να στηρίξει ε, την προσπάθεια για απάλληφη της ενεργειακής ένδυας. ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, σίγουρα αυτή είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, νομίζω στο πλαίσιο της ε, οδηγίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Κυρία Κάπελ, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe, είναι πολύ σημαντική και εμείς έχουμε την ίδια άποψη. Χρειάζεται ισχυρή, ε, χρειάζονται ισχυρές υποδομές έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα. Υπάρχει και το παράδειγμα της αιωλικής ενέργειας στη Βόρεια Γερμανία, όπου παράγονται πλεονάσματα ενέργειας. Και το θέμα είναι το πώς αυτό το πλεόνασμα θα πάει στα βιομηχανικά κέντρα του Νότου, αλλά και στους ε, καταναλωτές. Το θέμα είναι η έλλειψη υποδομών. Και εδώ το Connecting Europe θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Τώρα, ο κατάλογος PCI. Δεν υπάρχει θέση επίσημη από την Αυστριακή Προεδρία, διότι θέλουμε πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχτούν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Κύριε Φρόιντ, με ρωτήσατε την άποψή μου για τον ΙΤΕΡ, Να αντιδραστήρα αυτό. Η πυρηνική σύνδεξη είναι κάτι που θυμάμαι μόνο από το μάθημα της φυσικής στο σχολείο. Ίσως ε, για μένα πάει δεκαετίες πίσω, μάλλον και για σας. Ίσως θα θυμάστε πόσο συναρπασμένος ήταν ε, ο δάσκαλος, ο φυσικός μας από τις ε, δυνατότητες που έχει η πυρηνική σύνδεξη. και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε διάφορους τομείς ε, τις δυνατότητες που μας παρέχει. Χρειάζεται λοιπόν ε, να δώσουμε έμφαση στην έρευνα. Βέβαια, μας είπατε πως πρέπει να είμαστε και αξιόπιστοι σε αυτά που λέμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρότασή μας, την οποία έχουμε ήδη εγκρίνει για το 2030 είναι πολύ φιλόδοξη. Έχουμε στόχο λοιπόν το 50-55% της συνολικής μας ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες και έχουμε στόχο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι και 100% ανανεώσιμη ενέργεια, να γίνουμε ενεργειακά αυτάρκης δηλαδή. Να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό αν θέλετε, εισαγωγές-εξαγωγές. 36% μείωση διοξιδίου του άνθρακα. Οι στόχοι μας είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και ίσως ε, όταν ξανασυναντηθούμε σε μερικά χρόνια θα με ξαναρωτήσετε έτσι με διάθεση επικριτική αν έχουμε καταφέρει αυτούς τους στόχους. Κύριε Μπούζεκ, γραμμές διασύνδεσης, η ερώτησή σας αφορούσε αυτό. Φυσικά αυτό μας απασχολεί τι, ε, τι είναι ακριβώς αυτή η γραμμή διασύνδεσης, το interconnector. Πρέπει να καταλήξουμε σε έναν ορισμό, σίγουρα. Όμως δεν είμαστε ακόμα σίγουροι εάν αυτός ο ορισμός ε, θα πρέπει να είναι 100% εναρμονισμένος με εκείνον που, στον οποίο αναφέρεστε, για, που βρίσκεται στην οδηγία για, το αέριο. Ακόμα δεν έχουμε λοιπόν αποκρισταλλώσει τη θέση μας, όμως ε, σίγουρα ε, δεν τίθεται θέμα για το ότι πρέπει να καταλήξουμε σε έναν ορισμό. Αυτός λοιπόν, αυτός, λοιπόν ήταν ε, νομίζω και ο κατάλογος των ερωτήσεων. Νομίζω πως απάντησα σε όλους, οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και θα περιμένουμε την κυρία Κέστιγκερ. Ίσως και με το μωρό να έρθει, δεν ξέρω. And thank you very much for visit Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ladies and gentlemen, let us go ahead. Uh, Κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα το επόμενο σημείο της μερικής διαταξής μας. Επίσκεψη του Νόρμπερτ Χόφερ, Ομοσπονδιακού Υπουργού Μεταφορών, Καινοτομία και Τεχνολογίας της Αυστρίας. Υπέροχα, φανταστικά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Γιατί θέλουμε να δούμε το ένα θέμα μετά το άλλο. Πολύ σημαντικά θέματα αυτά για μας. Το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη και το πρόγραμμα για το διάστημα. Πιθανότατα. Στο παρελθόν δεν είχαμε ποτέ ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα για το διάστημα όπως αυτή τη φορά. Επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον και φυσικά συνεχίστηκε ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη. Θέλουμε ε, να Πάμε προ την ηλεκτρική ενέργεια, πολύ περισσότερο από ό,τι στο αέριο και έχουμε και συγκεκριμένε προτάσει εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν μπορούσα, κύριε Υπουργέ, να σα ζητήσω να ξεκινήσουμε με τη δική σα παρουσίαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Είχα και την ευκαιρία να ακούσω λιγάκι προηγουμένω που είχα μπει. Μιλήσατε για την ενεργειακή ασφάλεια. Πολύ ενδιαφέρον θέμα που δείχνει επίση το πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να συνεργαστεί σε ουσιαστικούς τομείς. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε και αυτές μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μόνο από κοινού. Είμαστε, ζούμε τη μια εποχή των μεγάλων προκλήσεων, των μεγάλων αλλαγών. Εμείς ε, τώρα έχουμε την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι είναι καθήκον μιας υπεύθυνης προεδρίας αφενός να συμβάλλει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βιώσει ένα αισιόδοξο μέλλον. Από την άλλη όμως την Προεδρία να την ασκήσουμε προσεκτικά έτσι ώστε αυτά που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα να διαφλαχθούν. Στόχοι είναι ειρήνη διαρκείας, ελευθερία και ευημερία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές εξάλλου και οι ιδέες των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκέφτηκαν ε, να μεριμνήσουν για μια ε, καλή οικονομική συνεργασία. Ε, μια συνεργασία που είχε υποφέρει λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν από αυτόν. Μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Στην Ευρώπη διασφαλίζεται η ελευθερία και η ειρήνη. Τώρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Κύριο πρόβλημα είναι ο εντονότερος, η εντονότερος, ανταγωνισμός. Ε, αν δούμε λιγάκι τις εξελίξεις στον κόσμο, νομίζω ότι ο πρόεδρος κύριος Τραμπ θα έρθει σήμερα το βράδυ εδώ ε, και ο ίδιος επιδιώκει τον προστατευτισμό Βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε τελικά πόσο πολύ θα φυγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτόν τον προστατευτισμό. Όμως θα φυγεί. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη Ρωσία, έχουμε την Κίνα ε, που αναπτύσσεται πάρα πολύ και η Κίνα τι κάνει, κάνει και περιοδία για να αγοράσει, να αγοράσει λιμάνια και πολλά άλλα διαστημική τεχνολογία. Έχουμε και την Ινδία και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμεθα λοιπόν να δεχτούμε ότι τα κράτη-μέλη μόνο τους ε, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνεργασία. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι σε αυτή τη συνεργασία ε, και τα σώματα υπέρ του ανταγωνισμού και της ε, διαφύλαξης της Ευρώπης ως έδρα επιχειρήσεων. Μας ενδιαφέρει επίσης και η κλιματική αλλαγή. Ευτυχώς έχουμε το πρόγραμμα Κοπέρνικος που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρξουν αποτελεσματικά μέτρα για βιώσιμη ανάπτυξη και υπάρχουν κίνδυνοι από ακραίες τάσεις, ε, υπάρχει τρομοκρατία. Αν λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις, κατανοούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο δύσκολο και αν είναι. Καλούμεθα να επεξεργαστούμε κοινέ λύσεις και καλούμεθα να αναλάβουμε ευθύνη έναντι των πολιτών. Ξέρετε, το σύνθημα της ε, Προεδρίας μας είναι το ρομπότ προστατεύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να απομονωθεί. Επειδή θα μιλήσουμε και για θέματα του διαστήματος, ε, τίποτα δεν ενώνει τόσο πολύ όσο οι κοινοί στόχοι. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να πλησιάσουμε περισσότερο τον πολίτη, το να σταθεροποιηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών ε, ε, στις διαπραγματευτικές ικανότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι και στις δικές σας τις χώρες γίνονται σφιγμομετρήσεις και ρωτούν τους πολίτες σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε την Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω εμείς ε, ως πολιτικοί οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και πολύ συχνά υποπίπτουμε στο λάθος ότι οποτεδήποτε εμφανίζονται αδυναμίες στην πολιτική των κρατών μελών, τα κράτη προσπαθούν να μετακυλήσουν το βάρος σε άλλα κράτη. Ως εκ τούτου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πούμε αν κάτι δεν πάει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν φταίνε αυτοί εκεί πάνω, αλλά την ευθύνη τη φέρουμε εμείς, γιατί και εμείς όλοι μας είμαστε ε, εκείνοι που στέλνουμε τους ε, πολιτικούς και εκλέγουμε πολιτικούς στα κράτη-μέλη. Και ελπίζω ε, και αυτό να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου κατά τους επόμενους έξι μήνες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να απαντήσουμε στα προβλήματα των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκπρόσωπος, υψώνει την φωνή των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο θεσμός εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Άρα φέρει και άμεσα την ευθύνη. Εσείς είστε εκείνοι που θα λογοδοτήσετε ε, στους ε, πολίτες όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ισχυρός εταίρος, απολύτως απαραίτητος για την επίτευξη των κοινών στόχων. Για μας, ε, για την Προεδρία μας, το Κοινοβούλιο είναι και ένας ιδιαίτερα ε, σημαντικός συνδετικός κρίκος. Κυρίε και κύριοι, αυτή είναι η βασική μας στόχη. Από αυτούς ξεκινάμε και τώρα θα αναφερθώ σε θέματα που αφορούν στο διάστημα. Να σας πω πόσο σημαντικό είναι το θέμα του διαστήματος για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το τομέα, στο τομέα του διαστήματος, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ε, στρατηγική, μια στρατηγική σημασία. Έχουμε τα προγράμματα Κοπέρνικους και Γαλιλαίος σε ψηλό επίπεδο και εκεί ε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρυβόμαστε σε σύγκριση με άλλες ε, διαστημικές χώρες. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Έχουμε λάβει ευφυείς αποφάσεις, έχουμε σαφείς στόχους. Έχουμε 22 δορυφόρους για το πρόγραμμα Γαλιλαίος. Αυτοί βρίσκονται σε τροχιά διαστήματος και αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρειαζόμαστε προφανώς το δικό μας το σύστημα. Η δορυφορική πλοήγηση μας ακολουθεί κάθε μέρα. Το σύστημα πλοήγησης, το GPS, το ξέρουν και τα παιδάκια. Ε, έχουμε πολύ καλή σχέση βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αν δεν υπήρχε πια αυτή η ασφάλεια, ξέρετε ότι με το GPS ε, μπορώ, μπορώ ανα πάσα ώρα και στιγμή να επιφέρω αλλαγέ, να κλείσω το σύστημα. Και κάποιος που οδηγεί, μπορεί να του είναι δυσάρεστο, ή για τον πιλότο ε, που οδηγεί με σύστημα GPS. Τα παλιά συστήματα χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο. Τα GPS χρησιμοποιούν πλέον οι πιλότοι. Υπάρχουν ε, και συστήματα προσγείωσης με GPS. Αυτοί οι πιλότοι εξαρτώνται, εξαρτώνται απόλυτα από το σύστημα GPS. Αν λοιπόν αλλάξει κάτι, αν ε, προκύψουν άλλα συστήματα, καταλαβαίνετε ότι υφίσταται ένα σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, ε, τις υποδομές πρέπει να τις εξασφαλίσουμε, τεχνικά πρέπει να βελτιωθούμε και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η χρήση διαστημικής ε, τεχνολογίας στον τομέα της προστασίας του κλίματος, της αηφόρου ανάπτυξης ε, και η πλοήγηση ε, παίζει απίστευτα σημαντικό ρόλο. Η διασφάλιση αποτελεσματικής governance για το διάστημα είναι πολύ σημαντική. Ενίσχυση των συνεργειών και με άλλα προγράμματα αυτά είναι στόχος της Αυστριακής Προεδρίας. Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σε αλλαγές που προκύπτουν στον τομέα του διαστήματος. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις όπως την εμπορευματοποίηση του New Space, να αντιμετωπίσουμε και τα πόβλητα του διαστήματος γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα, ας πούμε, στέλνονται οχήματα στο διάστημα. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, στις 30 Νοεμβρίου, σε επίπεδο υπουργών, θα έχουμε μια σχετική συζήτηση και εκεί θα συζητηθούν κάποια σημαντικά θέματα του μελλοντικού διαστημικού προγράμματος. 5 και 6 Νοεμβρίου ε, διάσκεψη ε, για το διάστημα στο Γκράτς. Ο κύριος Σαλίνη είναι ο εισηγητής. Ελπίζω να έρθει στο Γκράτς ο κύριος Σαλίνη και θέλω να υπογραμμίσω και τη συνεργασία μας με την Ισπανία. Όλα αυτά για μας είναι πολύ σημαντικά. Και τέλος, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να αναφερθώ σύντομα ε, στο, σε, ένα θέμα, το, σε ένα θέμα top level, domain, αυτό έχει να επιδείξει μόνο επιτυχίες. Είναι ιδιαίτερα προσφυλές ε, στους ε, Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Είναι θέμα ευρωπαϊκής ταυτότητας στο διαδίκτυο. Εμείς ε, συμφωνούμε πρέπει να εξυγχρονιστεί το domain, το EU domain και χαιρετίζουμε να υπάρχει ένα φόρουμ multi-stake η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερωτάται για αυτό το EU domain και θέλουμε να επιτύχουμε την συμμετοχή του Συμβουλίου διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ε, μάλιστα, ίσως μπορούμε να κάνουμε και κάποια περισσότερα. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εμφερθήκατε σε αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο για το μηχανισμό Συνδέτης στην Ευρώπη και το πρόγραμμα του διαστήματος. Ο κύριος Κάριν, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Χόφερ που ήρθε στο Κοινοβούλιο. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον, ε, είναι πολύ σημαντικό στο τομέα των μεταφορών. Πολύ σωστά είπατε, η ε, αεροπλοεία αλλά και οι οδικές μεταφορές, τα διόδια, όλα αυτά συνδέονται και στα πλαίσια του Connecting Europe θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, ακριβώς όπως η εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών θα και η εσωτερική αγορά ενέργειας ε, είναι πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Βέβαια, οι φυστάμενες δομές έχουν λίγο πολύ οδηγήσει σε ολιγοπόλια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Ωστόσο, νομίζω πως η προσέγγιση σας είναι σωστή, διότι ε, αν καταφέρουμε να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες το 100% τότε το 100% των πολιτών θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται όμως ε, να δράσουμε εγκαίρω και σωστά έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους καταναλωτέ και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια. Τώρα, το Connecting Europe ε, Νομίζω πως είναι το κατάλληλο πλαίσιο για το διαστημικό πρόγραμμα, αλλά τι γίνεται με, την, ε, με τις ε, συνδέσεις. Σίγουρα είναι μια καλή πλατφόρμα επικοινωνίας. Ε, επίσης ε, βρίσκεται σε, έχει καλή συνεργασία με το ΣΤΟΑ, την Υπηρεσία του Κοινοβουλίου για τις Τεχνικές Μελέτες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια παράκληση. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οργανισμοί οι θεσμοί αυτοί να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, διότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι υποδομές επικοινωνίας θα είναι κέρια σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μέλλον, αλλά ήδη από τώρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αντικαθιστώ τον συναδελφό του που Είναι αρμόδιος ε, για το θέμα αυτό, αλλά έπρεπε να μεταβεί στην Πράγα. Επομένως, ε, τον αντικαθιστώ εγώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε στην αρχή της ομιλίας σας. Μιλήσατε για προστατευτισμό και για την απειλή αυτή. Όπως ξέρετε, υπάρχουν προστατευτικές τάσεις εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο εκτός. Παραδείγματος χάρη, αυτή η ιστορία να προσπαθήσουν κάποιοι να θέσουν εμπόδια στην ε, κεντρική Ευρώπη. Εμείς το έχουμε συζητήσει αυτό επανειλημμένως και ελπίζω τελικά οι χώρες της περιοχής μας ε, να βοηθηθούν από την Προεδρία σας, γιατί εμείς έχουμε πολλές ελπίδες στη δική σας Προεδρία. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσετε να θεωρείτε και τη δική σας χώρα, χώρα της ε, Κεντρικής Ευρώπης, όπως κάνατε τη δεκαετία του 80. Θέλω να ρωτήσω τώρα, τι στόχους έχει θέσει η Αυστρική Προεδρία σε ό,τι αφορά το διαστημικό πρόγραμμα πότε θα το υλοποιήσετε και ποια χρονική στιγμή. Πιστεύετε ότι πριν τις ευρωεκλογές του 2019 μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ Συνομβουλίου και Κοινοβουλίου, γιατί φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα εργαστεί η Προεδρία σας στο Συμβούλιο. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το τι σκέφτεται η δική μας πολιτική ε, ομάδα, η Τόρις, η συντηρητική από τη Βρετανία. Αν ε, θα συμμετάσχουν οι Βρετανοί σε αυτά τα προγράμματα, όπως το Γαλιλαίο, το χάρη, θα μας φαινόταν πολύ θετικό. Γιατί θα ήταν θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν μετά το Brexit θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως το Γαλιλαίο. Εσείς τι πιστεύετε και τι πιστεύει η Αυστρική Προεδρία για το θέμα αυτό. Εκ μέρους του ΙΕΝΕΦ. E η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Χόφερ, χαίρομαι πολύ που σας καλωσορίζω σήμερα στην Επιτροπή μας. Να σταθώ λίγο σε, αυτό, σε αυτή την παγκόσμια διάσταση στην Επιτροπή μας. Ε, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε, και ε, στον τομέα της ε, ψηφιοποίησης. Πρόσφατα είδαμε μία μελέτη του ελεκτικού συνεδρίου σύμφωνα με την οποία χρειάζεται πιο γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση στην Ευρώπη. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψει σε ό,τι αφορά την ευρυζωνικότητα, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Η Ήπεθρο εξαρτάται απόλυτα από την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητα, ενώ αντίθετα στις ε, πόλεις υπάρχει μεν ε, αφ αυτό όμως δεν προβλέπεται ε, περαιτέρω ανάπτυξη στη στρατηγική για μετά το 2020. Υπάρχουν σχέδια με τα οποία χρειάζονται όμως ε, επικαιροποίηση, επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επεξεργαστεί εκ νέου την οδηγία για τις ε, δημόσιες συμβάσεις και επίσης το ΕΦΣΙ και το Connecting Europe θα συμμετέχουν στην χρηματοδότηση μικρότερων ε, σε έργων. Χρειάζεται όμως να στηριχθεί η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη. Έπειτα, διάστημα, διαστημική βιομηχανία και οικονομία. Στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, υπάρχει καταρχάς ε, με χρηματοδότηση 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για το νέο διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης. Ε, είπατε κι εσείς τα, προγράμματα, τα συστήματα Γαλιλαίο, Κοπέρνικος που θα αποτελέσουν συστατικά στοιχεία στο νέο πλέγμα σχετικά με την ασφάλεια. Είπατε επίση ότι για την Αυστριακή Προεδρία η πολιτική του διαστήματος είναι σημαντική, αλλά νομίζω πως δεν γίνονται αρκετές προσπάθειες να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα να σας ζητήσω να δώσετε απαντήσει και να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις βάσει τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ε, τέτοιο το θέμα τι θα κάνουμε με το θέμα της ε, το θέμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών ε, επιτέθηκε συμβαστική πρόταση αλλά αυτή είναι καλή συμβαστική πρόταση και νομίζω ότι Είμαστε ικανοποιημένοι. Δεσπά, εγώ είμαι ικανοποιημένο και φαντάζομαι ότι και εσείς ε, είστε ικανοποιημένο. Θίξατε το θέμα της ε, επικοινωνίας ε, στο διάστημα των εξωτερικών οργανισμών, των θεσμών που υπάρχουν σχετικά με αυτή την επικοινωνία στο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Παράλληλα όμως χρειαζόμαστε και ε, σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν πάρα πολλές επικαλύψεις, δυστυχώς αυτό και τις τελευταίες ημέρες πολλοί μου είπαν «Ξέρετε, χρειαζόμαστε μία σαφή γραμμή να ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος γιατί». Και είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι στο πλαίσιο αυτής της Προεδρίας αποκοινούμε το Κοινοβούλιο και αποκοινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρούμε ικανοποιητικέ λύσεις. Ο κύριος Τουστανόφσκι μίλησε για τον προστατευτισμό που μας συνοδεύει όχι μόνο όσον αφορά στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά είπε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να πω κάτι πολύ προσωπικό. Εγώ μεγάλωσα στο ανατολικό κομμάτι της Αυστρίας, πίσω από το Σιδηρούν παραπέτασμα. Όταν λοιπόν πέφτει αυτό το, όταν πέφτει το παραπέτασμα και βεβαίως βλέπει κανείς πως έχει προχωρήσει η πρόοδος, εμείς εκμεταλλευτήκαμε πάρα πολύ το ότι έπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα. Και βλέπουμε πόσο ε, στενή σχέση ανάμεσα στους πολίτες του δικού μου κρατηδίου και τους ε, συμπολίτες μας ε, στην Ουγγαρία. Έχουμε λοιπόν έναν κοινό δρόμο ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω κανένα. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, παρορμητικά να ε, αποφαινόμεθα για τάσεις για εξελίξεις και να κόβουμε και τη συζήτηση. Θεωρώ ότι η διπλωματία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ η διπλωματία καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και νομίζω ότι είναι ένα του της Αυστρίας τα πάει πολύ καλά με τη διπλωματία. Και επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Πραγματικά έχουμε μια πολύ καλά λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Και αυτός είναι και ένα λόγος γιατί το Συμβούλιο Υπουργών θα τα πάει πολύ καλά. Όχι γιατί υπουργοί είναι μεγαλοφίε, κάθε άλλο. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι σύμβολοι, οι οποίοι προσπαθούν να αναζητήσουν ε, συμβασμού λύσει. Εμείς λοιπόν, λοιπόν οι υπουργοί έχουμε τη χαρά να ανακοινώνουμε το ευχάριστο μήνυμα. Αλλά η προεργασία γίνεται από άλλου. Ε, οι συζητήσει λοιπόν έχουν ήδη ξεκινήσει ε, και βαδίζουν πολύ καλά. Η Αυστρία, σα λέω, θέλει να είναι γεφυροποιό. Κατά πόσον θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ε, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Αλλά εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε το εφικτό κάνατε μία ερώτηση σχετικά με το Brexit, τι θα γίνει με το πρόγραμμα Γαλιλαίος, πώς θα επηρεάσει το Brexit το πρόγραμμα αυτό. Ξέρετε, σε τελική ανάλυση πρέπει να ασχοληθούμε με το πακέτο στο σύνολό του και να βάλουμε ε, το Γαλιλαίο, το πρόγραμμα αυτό με, σε συνδυασμό με το Brexit, εγώ πιστεύω ότι τελικά ε, θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό. Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες αλλαγέ σε προσωπικό επίπεδο. Η κυρία Δόκτωρ Κάπελ ε, έθεσε το θέμα της ε, ψηφιοποίηση. Νομίζω ε, σήμερα είναι σημαντικό όχι μόνο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια και τίποτε άλλο, χρειαζόμαστε την ψηφιοποίηση ε, η ψηφιοποίηση είναι καθοριστική σημασία και όσον αφορά την επέκταση της ε, ευρυζωνικότητας πράγματι υπάρχουν νέες εξελίξεις δηλαδή το 5G Fiber to Home δεν θα είναι τόσο σημαντικό όσο τώρα δεν πρέπει οι οπτικές ίνες να φτάσουν σε κάθε σπίτι, αλλά κάθε σπίτι πρέπει να έχει ευρυζωνικότητα. Μία στρατηγική δηλαδή που ε, θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει απόλυτο συντονισμός ανάμεσα στις οπτικές ίνες και, τα, και την τεχνολογία 5G. Και αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε για όλες σας τις παρατηρήσεις και για την εναρκτήρια ομιλία σας. Και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Πάμε στο επόμενο σημείο. Το 26. Έχουμε την εσωτερική αγορά για την ηλεκτρική ενέργεια, αναδιατύπωση του κανονισμού και κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά στην ηλεκτρική ενέργεια. Αναδιατύπωση, οδηγία. Ο κύριος Κάρινς είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Σε κάτω από τρία λεπτά και μάλιστα σε κάτω από ένα λεπτό μπορώ να τα πω. Ολοκληρώσαμε την ε, ψηφοφορία μας ε, στην Ολομέλεια στις 28 Φεβρουαρίου και περιμέναμε πολύ καιρό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις υπό τη Βουλγαρική Προεδρία. Τελικά έγινε αυτό στα τέλη Ιουνίου. Ουσιαστικά είχαμε συνεργασία με την ε, επερχόμενη Αυστριακή Προεδρία. Είδαμε και από τις δύο πλευρές ποιες ήταν οι πολιτικές προκλήσεις που συνδέονταν με τεχνικές ε, ε, τεχνικά θέματα που θα λάβουν χώρα, θα συζητηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου και στις 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τριμερή διάλογο. Έτσι λοιπόν ξεκινά επιτέλους η όλη δουλειά και έχουμε να αποθέσει τις ε, ελπίδες μας στην Αυστριακή Προεδρία για να ολοκληρωθεί ο φάκελος αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας τους. Μάλιστα, είναι όλα σαφή πιστεύω, αλλά αν θέλει κάποιο να θέσει κάποια ερώτηση, να κάνει κάποια παρατήρηση, ωραία, σας ευχαριστώ. Γιατί πριν δύο εβδομάδες αρχίσαμε τη συζήτηση, δεν θα είναι εύκολη. Και ο επόμενος τριμερής διάλογος είναι για το Δεκέμβριο. Μάλιστα, ευχαριστώ λοιπόν για την ε, παρουσίασή σου. Λοιπόν, 28 και 29 από κοινού. Πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματο Πλησίωρευση Καινοτομία Ορίζων Ευρώπη το κανόνα συμμετοχή και διαδοσή του. Και δεύτερο θέμα πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματο υλοποίηση του προγράμματο Ορίζων Ευρώπη. Πρόγραμμα πλαίσιο έρευνα και κοινοτομία. Δύο θέματα έχουμε εδώ και δύο εισηγητέ τον κύριο Ντανίκα και τον κύριο Κριστιαν Έλλερ. Παρακαλώ, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψε για αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο. Ο κύριος Ντανίκα, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, όσους αυτό το μήνα ήταν δίπλα μου και με βοήθησαν να παρουσιάσω και να ετοιμάσω μία αξιοπρεπή έκθεση και ευχαριστώ όλους που έκαναν την προσπάθεια να είναι δίπλα μου και να κατανοήσουν τι έκανα. Γιατί βρίσκονται εδώ ακόμη. Επίσης, οι συνάδελφοι από την Ήτρε συμμετείχαν. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν και τέλος την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνεχώς προσπάθησε να είναι παρούσα και να συνεισφέρει. Διατηρώντας την αρχική υπόσχεση, δηλαδή να παραδοθεί η έκθεση αυτή την εβδομάδα, οργάνωσα και δύο διασκέψεις και πολλές άλλες διμερείς συναντήσεις όπου προσπάθησα να λάβω feedback από τους κύριους πρωταγωνιστές στον τομέα της έρευνας και της κοινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλαβαίνω αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Για ποιο λόγο και πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά καλύτερα για το μελλοντικό πρόγραμμα Ευρώπη, Horizon Ευρώπη και για το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ήθελα να αναφέρω τα κύρια σημεία. Ήδη έχουμε στην κατοχή μας σήμερα μία εκδοχή της έκθεσης της 10 Ιουλίου και θα προσπαθήσω να στείλω το σχέδιο της έκθεσης αυτής, ε, στο στάδιο που βρίσκεται, να δούμε ποια είναι η δυναμική της έκθεσης αυτής. Έτσι λοιπόν, θα αναφέρω κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα τα κυρία σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά την αύξηση του προπολογισμού 20 δισεκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές. Στην πρόταση της Επιτροπής υπάρχει μία πρόταση προϋπολογισμού σε τρέχουσε τιμέ ε, μόνο για 83 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε προσθήκη μόνο 1,4 δισεκατομμύρια σε τρέχουσε τιμέ. Η υποστήριξή μας έχει εκφραστεί ήδη για να έχουμε 20 δισεκατομμύρια σε τρέχουσε τιμε Σημείο 2. Η ενδυνάμωση της ε, έρευνας ε, είναι κάτι σημαντικό, κυρίως γιατί η θεμελιώδης έρευνα είναι ένας ε, πολύ σημαντικός τομέας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τρίτο σημείο είναι η εισαγωγή της αρχής της αμοιβαιότητας. Θα πρέπει να προσαφηνίσουμε όλη αυτή την κατάσταση γιατί δυστυχώς από όλα όσα είδα η κατάσταση είναι κάπως περίεργη. Απ' τη μία, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να μπορούν να κατεναμηθούν σε project που είναι πολύ καλής ποιότητας και που προτίζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά χρήματα, δυστυχώς δεν έχω νούμερο να σας πω, που ε, ε, περισσεύουν αυτή τη στιγμή από τον ορίζοντα 2020. Τώρα, τώρα πόσα χρήματα δόθηκαν και για τις συνδεδεμένες χώρες αλλά και για τις τρίτες χώρες αλλά πιστεύω ότι η αρχή της αμοιβαιότητας είναι κάτι υποχρεωτικό γιατί θα ήταν δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί δεν δίνουμε σε κάποιον πρόσβαση σε πόρους που είναι χρήματα των Ευρώπων φορολογουμένων και οι οντότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, θα είχαν δικαίωμα πρόσβασης ε, σε προγράμματα και project που έχουν χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο κράτος. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Ένα άλλο σημείο που εντόπισα και θα ήθελα να το αποσαφηνίσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης είναι το θέμα των κανόνων διανοητικής ιδιοκτησίας γιατί υπάρχει, για να υπάρχει ουσιαστικά ε, μία αποτίμηση της αξίας της ευρωπαϊκής έρευνας. Οι νέοι συμμετέχοντες και οι μικροί χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται στήριξη και συμβουλές για να ξέρουν πώς θα προστατεύσουν καλύτερα τα διανοητικά τους δικαιώματα και ταυτόχρονα ξέρουμε με μεγάλη ακρίβεια ποιος έχει τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέμπτο σημείο που θέλω να εισαγάγω στο πλαίσιο της εκθέση αυτής αφορά την ε, πρώτη εμπορική εκμετάλλευση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα που θα έχουν χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να υπάρχει, για να υπάρχει μεγιστοποίηση του αντικτύπου αφενό και αφετέρου, πρόσθετη αξία, προσθεμένη αξία των ε, δαπανών που προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι λοιπόν, αυτό το θέμα, η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να σας πω πολύ γρήγορα οι συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα δούμε με τους συναδέλφους από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Θα έχουμε σημεία αριστείας και επίσης θέλουμε ε, και ίσες πληρωμές, ίσους μισθούς για ίση εργασία. Δηλαδή έχουμε συζητήσει, παραδείγματο χάρη, δίκαιους μισθούς για τους οδηγούς φορτηγών. Εγώ νομίζω ότι και εδώ, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται για τους ερευνητέ ε, οι οποίοι εργάζονται σε συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα. Θα, μία αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει βάση της αριστείας, όχι βάση του φύλου ή άλλων κριτηρίων. Και η ε, μείωση του χάσματος στον τομέα της έρευνας ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και καλύτερη ανταλλαγή ε, της αριστείας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά είναι τα δέκα σημεία που ήθελα να αναφέρω και αυτό είναι το έγγραφο το οποίο θα δώσω και στη γραμματεία προκειμένου να προσαρτηθεί στην έκθεση έτσι όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Και πάλι σας ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σύντομοι, να είμαστε γρήγοροι, γιατί έχουμε προθεσμία για τη μετάφραση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ναι, αυτή την Παρασκευή η έκθεσή μου θα πάει για μετάφραση. Θα τη δώσω στη γραμματεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Έλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ντανίκα. Νομίζω πως υπάρχει αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση. Θέλαμε η θέση που, στην οποία θα καταλήξουμε να είναι συνεκτική. Αλλά αυτό ήταν το γενικότερο κλίμα και με όλους τους σκιώδεις. Τώρα, Επί τούτου, νομίζω πω αυξάνεται ο γενικότερο προπολογισμό κατά 120 δισεκατομμύρια. Επιμένω όμω, δεν είναι αύξηση αυτή του προπολογισμού, απλά αντικατοπτρίζουμε και εμεί αυτά που αποφασίστηκαν από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων για την γραμμή του προπολογισμού που θα είναι αφαιρεμένη στην έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε το Συμβούλιο να ε, ακολουθήσει τι ε, δικές του που έλαβε πριν από 10 χρόνια. Τώρα, στον πρώτο πυλώνα θα θέλαμε περισσότερη έμφαση στο proof of concept. Επίση, η σφραγίδα αριστεία ε, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να δοθεί περισσότερη έμφαση στους νέους ερευνητέ. Τώρα, το πρόγραμμα Marie Curie θα πρέπει να ε, φροντίσει θέματα ισότητας ε, των φύλων, όχι απλά να το αναφέρουμε αλλά να βοηθάμε τις γυναίκες ερευνήτρες. Ε, επίσης, ως προς το πρώτο πυλώνα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ή στρατηγική σε υποδομές ε, στα λιγότερα αναπτυγμένα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, σε θέματα χρηματοδότησης από το ΕΦΣΥ, από θέματα χρήσης του Open Science Cloud, το συζητούσαμε εδώ και πολλά χρόνια, να είχαμε ένα τύπου υπολογιστικό νέφος με ανοιχτό χαρακτήρα, το οποίο επίσης θα ε, ασχολούταν και με επιστημονικά θέματα, ερευνητικά, μετά ομάδα για τις ε, κοινωνίες χωρίς αποκλεισμό. Αυτό ε, θα χωριστεί στα δύο διότι με την παρούσα μορφή του έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα. Επίσης, νομίζω είναι αυτονόητο πως υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό. Ναι, αναφερόμαστε σε σχεδιασμό με πιο στρατηγικό χαρακτήρα, πιο ανοιχτό κτλ. Από την άλλη όμως ε, πρέπει να εντοπίσουμε τα προβληματικά σημεία, να δούμε ποιο είναι το, ποια είναι η αποστολή μας, το έργο μας, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Θέλουμε να περιορίσουμε λίγο εδώ την κατάσταση, το πεδίο εφαρμογή και γι' αυτό χρειάζεται ορισμός. Τώρα για τις ε, εταιρικέ σχέσεις πρέπει να δούμε τις συνέργειες, τη συνεργασία και τη μόγλευση της ε, Βιομηχανία, ε, προγράμματα όπως ο καθαρός ουρανός είναι πάρα πολύ σημαντικά, θέλουμε να παραμείνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το EIT, δίνεται έμφαση σε αυτό. Θέλουμε να ε, κρατήσουμε τα πλεονεκτήματα. Ε, για, τη, τα KICS, να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση αποστολές τώρα, όπως ε, είπα ήδη και για την πρόταση για το στρατηγικό σχεδιασμό, θέλουμε να μειωθούν οι αποστολές ε, στον πρώτο στο πρώτο στάδιο στρατηγικού σχεδιασμού, ακριβώ γιατί όταν υπάρχουν 50 αποστολέ, ε, χάνεται η ουσία, χάνεται η έμφαση. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια σαφέστερη κατεύθυνση του προπολογισμού εκεί. Προσανατολισμός λοιπόν στις παγκόσμιες προκλήσεις. Επίσης, ε, συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα, με ερευνητικά, με ε, συνεργασίες. Η έρευνα δεν είναι κάτι αυτόνομο. Πρέπει νομίζω να βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα και τη σχέση της ε, με την βιομηχανία. Νομίζω πως πρέπει να μειωθεί προϋπολογισμός για τις αποστολές σε πρώτο στάδιο να, υπάρχει, να υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλογής και όχι απλά να χρηματοδοτούμε έτσι στα τυφλά αποστολέ οι οποίες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Θέλουμε πιο γρήγορη διαδικασία από τη βάση προ την κορυφή, θέλουμε να επεκτείνουμε το, τα πιλωτικά project από τον ορίζοντα 2020 και σε ομάδες προγραμμάτων και επίσης θέλουμε να επιταχύνουμε την διαδικασία, να υπάρχει ένα χρονικό όριο έξι μηνών για την ε, για ε, χορηγήση χρηματοδότησης. Θέλουμε επίσης νέες πρωτοβουλίες αριστείας για τα λιγότερα αναπτυγμένα κράτη, έτσι αυτά να μπορούν να ζητήσουν ε, διεθνή χρηματοδότηση και να εκτελέσουν μεταρρυθμίσεις. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε πως η καλύτερη διαχείριση των δεδομένων είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με τις υποδομές αλλά και με το ανοιχτό επιστημονικό υπολογιστικό νέφος και το Heritage Cloud. Μετά πρέπει να διευρυνθούν να διευρυνθούν οι σφαγηδαριστές και σε άλλα προγράμματα, να συζητηθούν προτεραιότητες ε, θεματικές, για παράδειγμα ε, δημιουργικές βιομηχανίες, στήριξή τους, ε, στήριξη ε, της βιομηχανίας όχι μόνο όμως σε θέματα ενέργειας αλλά και σε άλλα θέματα υγείας, σπάνιες ασθένειες, παιδικός καρκίνος. Αυτό φυσικά είναι νομίζω άμεσα κατανοητό από τον απλό πολίτη, παραγωγή τροφίμων, κλιματική αλλαγή. Λίγη περισσότερη έμφαση δηλαδή σε ορισμένες θεματικές προτεραιότητες. Επίσης, να διευρύνουμε λίγο τον οριζοντά μας. Πρέπει να δούμε τη σύνδεση με τα διαρθρωτικά ταμεία, αυτό το 5%. Αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Δύο προτάσεις οι οποίες ήταν ο καθέφτης η μία της άλλης. Τώρα υπάρχει λίγο διαφορετική νομοθετική πρόταση, αυτή μετά, συνέργειε με, το, με τη Δημιουργική Ευρώπη δεν αναφέρεται καθόλου στην πρόταση. Πρέπει να δούμε τα χρηματοδοτικά μέσα, ακριβώ διότι θέλουμε να κρατήσουμε την ευελιξία. Στα νέα προγράμματα δεν υπάρχει δηλαδή μία λύση για όλους, αλλά έτσι λίγο πιο εξατομικευμένη είναι η προσέγγιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης πρέπει να είμαστε ειλικρινεί πως πρέπει να συζητήσουμε από την αρχή με πιο γενικούς όρους, διότι στον τρίτο πυλώνα του προγράμματος βλέπουμε ότι υπάρχουν τα πιο προβληματικά σημεία αλλά και τα πιο σημαντικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και ζητώ συγγνώμη που αναφέρομαι έτσι επιγραμματικά και τόσο γρήγορα σε αυτά, όμως ε, βιάζομαι να τελειώσω την έκθεση, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να την έχω υποβάλει. Νομίζω όμως πως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο από αυτά που ακούμε από τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, βλέπω ότι η θέση που θα, στην οποία θα καταλήξουμε απέναντι στο Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και τέλος, μια παράκληση προς το Συμβούλιο την τελευταία φορά 18 μήνες διαπραγματευόμασταν. Τώρα είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι, πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα, να ε, δώσουμε ασφάλεια στους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Όσο πιο φιλόδοξοι είμαστε, τόσο πιο καλά πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί έρχεται το 2020 το νέο πρόγραμμα και δεν θα είναι η πολιτική κατάσταση όπως τώρα, θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η καινοτομία θα έχει λάβει διαφορετικές διαστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάμε πίσω ότι και το Συμβούλιο θα έχει τη δική του θέση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριο Έλερ μίλησε, πιστεύω, σας σκιώδης για το πρόγραμμα Ορίζοντας. Θα ήθελετε τώρα να πάρετε το λόγο και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το ειδικό πρόγραμμα. For the second program. Μπορείτε τώρα να πάρετε το λόγο για το δεύτερο πρόγραμμα. Dopo. Okay. Allora, completiamo Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το, ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των ομιλητών. κυρία Καμπέσον Ρουίς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους δύο συγητές για την ενημέρωση και για τις καινοτομίες. Όλα αυτά είναι σημαντικά και θετικά. Απλώς να τονίσω κάποιες ιδέες για την ε, βιομηχανία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ορίσουμε καλύτερα το ρόλο ε, ή το πώς εκπροσωπούνται οι ΜΜΕ. Νομίζω ότι δεν το βλέπουμε πολύ καλά. Ήταν πολύ σημαντικό το εργαλείο, το μέσο για τις ΜΜΕ στον ορίζοντα 2020. Τώρα, συνεργίες. Αυτό το πρόγραμμα ε, δεν μπορεί να μιλά μόνο για την αναγκαιότητα, για συνέργεια. Πρέπει να γίνει πραγματικότητα διαφορετικά. Αν δεν μάλλον ε, βρούμε τους κατάλληλους μηχανισμούς ε, που επιτρέπουν την αλληλοσυμπληρωματικότητα και τελικά τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, αυτά τα κονδύλια που σχετίζονται με το 2020, ε, μόνο τότε θα μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι συνέργειες. Επίσης, για την σφραγίδα της αριστείας είναι πάρα πολύ περιορισμένη χρήση της. Επίσης, πρέπει να βρούμε μηχανισμούς που να δίνουν κίνητρα της πραγματικής συμμετοχής στις συνέργειες με άλλα ταμεία από την πλευρά των κρατών μελών. Πρώτος πυλώνας για την ανοιχτή επιστήμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο άνοιγμα και στο υπόλοιπο πρόγραμμα ίσως ε, θα έπρεπε να ε, υπάρχει ένα πολύ πιο ανοιχτό πρόγραμμα, όχι να επικεντρωθούμε μόνο στον πρώτο πυλώνα για τους νέους. Πολύ σημαντικό, μου φάνηκε πάρα πολύ θετική η πρόταση της Επιτροπής, συμπεριλαμβάνει και τις συνέργειες με το πρόγραμμα Εράσμους, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε προς ένα πολιτισμό που να προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους νέους χρειαζόμαστε και ένα πρόγραμμα ή ένα ειδικό μέσο που να μας επιτρέψει οι νέοι ερευνητές και οι πανεπιστημιακοί και οι διδακτορικοί να αποτελούν μέρος αυτού του προγράμματος. Επίσης, δυνατότητα αυτό να είναι ένα μέσο για να επιστρέψουν τα ταλέντα. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο, γιατί υπήρξε μια φυγή των ανθρώπων αυτών λόγω της οικονομικής κρίσης και κάτι ακόμη. Ο κύριος Νίκα Μα είπε ότι θέλει να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Πολύ καλό και αυτό. Απλώς θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα να μπορέσουμε να μετρήσουμε καλύτερα τον κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος, δηλαδή πόσο ωφελείται η κοινωνία από, αυτές ε, τις, από αυτά τα επιτεύγματα της επιστήμης ή κομισιόν. Στην πρότασή της έχει συμπεριλάβει δείκτες, μου φαίνεται σημαντικό αυτό, σημαντική καινοτομία και μπορούμε να εργαστούμε για τη βελτίωσή του, γιατί θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να φτάσει σε όλη την κοινωνία και να αποτελεί πραγματικά κινητήριο δύναμη τη αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε και επί του κοινωνικού αντικτύπου. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πάνω κάτω που σεβαστήκατε το χρόνο. Για το ECR, ο κύριο Καντονεύσκη. Ήρθε και η κυρία Κατσασενόφσκη. Αλήθεια δεν είναι. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δύο λόγια. Καταρχήν, Τσέχος συνάδελφος θέλει να πει στους ε, εισηγητές ε, ότι είναι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί εσείς ε, πραγματικά ανασηκώσετε τα μανίκια και αρχίσατε να δουλεύετε. Δύο-τρία πράγματα θέλω να τονίσω. Καταρχήν, υποστηρίζουμε τη θέση του κυρίου Νίκα, δηλαδή το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη να έχει μεγαλύτερο περιπολογισμό και να φτάσει στα 120 δις. Κάτι άλλο που μας φαίνεται πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία. Δηλαδή, όλες αυτές οι τροπολογίες που οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση για μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία, βεβαίως και θα τις υποστηρίξουμε. Είναι σημαντικό όταν διευρυνθεί αυτό το, το πρόγραμμα να υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι τροπολογίες ε, είναι απολύτως λογικές και θεμελιώδεις. Έτσι λοιπόν, ο εισηγητής από τη ΣΥΑΡ θα τις υποστηρίξει. Επίσης, υπάρχει το θέμα της ε, εξόδου του Brexit και στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο ορίζον Ευρώπη. Να δούμε τι θα συμβεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίρινγκ. Thank you, Chair. Um, about regulation uh, and... Ευχαριστώ για τους ε, κανόνες στη συμμετοχή στο Horizon Ευρώπη. Για το Horizon Ευρώπη έχουμε τον ίδιο στόχο να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική από τα σήμερα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη διάδοση της αριστείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διάφορων ταμείων, των διάφορων κονδυλίων. Το Horizon Ευρώπη θα πρέπει να έχει εναρμονισμένη προσέγγιση και ω προς ε, ε, το εντικό πρόγραμμα αλλά και τον κανονισμό. Ε, σε αυτό στοχεύουν οι δύο και τους υποστηρίζω πλήρως αυτό. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα ήθελα να ε, έχουμε κατά νου το πώς βλέπουμε τις μελλοντικέ εξελίξεις της έρευνας και κοινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιλογές που θα κάνουμε ως νομοθέτες θα έχουν επίπτωση ε, στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει έρευνα και αναπτύξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιπρόσθετα σε σχέση ε, με τι χώρε εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να έχουμε μία σχέση αμοιβαιότητα. Συνεπομονούμε να συνεργαστούμε κύριε Νίκα για το φάκελο αυτό μαζί σα. τώρα για το ειδικό πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Πιστεύω ότι η εστίαση θα πρέπει να γίνει στο πώς το ειδικό πρόγραμμα του Ορίζον Ευρώπη θα διαμορφωθεί. Όπως ε, είπε ο κύριο Έλερ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του προγράμματο για τους ερευνητές, όσους ε, προβαίνουν σε καινοτομίες ε, και του επενδυτέ. Μόνο έτσι μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνα. Έτσι λοιπόν, ανυπομονώ να συνεργαστώ και στο φάκελο αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο μαζί σα, κύριε Έλερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο, ο κύριος Νταλούντε. Thank you, Chair. So first... Ευχαριστώ. Καταρχήν για το πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ κυρία Νίκα για την πρόταση. Εκτιμούμε που εργαστήκατε τόσο γρήγορα για να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύουμε ότι η θέση σα να αυξηθεί ο προπολογισμό είναι ένα καλό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε για να προωθήσουμε καινοτομία και έρευνα ω τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ είναι βήμα προ την κατεύθυνση. Πρώτο σημείο. Είναι σημαντικό για μας ο ξερθολογισμός για το κλίμα να ενδυναμωθεί και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε μεγάλους καύσονες εξηρεσίες ε, ακόμη δεν ε, έχουμε μπει ε, στην πορεία να σεβαστούμε τους στόχους μας θα πρέπει να αυξηθούν τα μέσα γιατί θα αυξηθούν και οι προκλήσεις και επίσης θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να έχουν μια ευκαιρία να διακριθούν, να ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τεχνολογίες υψηλής ποιότητας. Είμαστε σκεπτικοί ως προς ε, την ιδέα της χρησιμοποίησης κονδυλίων από το Horizon Ευρώπη για γεωγραφικούς λόγους. Εμείς έχουμε διαφορετικά ταμεία για διαφορετικούς σκοπούς. Το, η αριστεία θα πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο για το οποίο επιλέγεται ένα project, ένα πρόγραμμα. Η εστίαση θα πρέπει να είναι στον αντίκτυπο όμως των προγραμμάτων. Αυτό είναι καλύτερο κριτήριο από τη γεωγραφία. Τρίτο σημείο. Ανησυχούμε για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και εμεί ω νομοθέτε αφήνουμε πολλά στην Κομισιόν. Εδώ θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να βρούμε λύσει που θα μα δώσουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Τέταρτο σημείο όλη η έρευνα και η καινοτομία βασίζεται στην ικανότητα των επιστημόνων, των Ινστιτούτων και των επιχειρήσεων και των πολιτών να έχουν ανοιχτή πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν τις επιστημονικές πληροφορίες και να αυξήσουν την εκμετάλλευση της γνώσης. Θα πρέπει να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσει πρέπει να ε, τεθεί και το θέμα ε, της διάστασης του φύλου. Θα πρέπει να έχουμε ίσους μισθούς για ισότιμη δουλειά. Για τον κύριο Έλερ τώρα, για το ειδικό πρόγραμμα, πρώτο σημείο. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι κλίματος και βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο και να είναι κύριο στοιχείο των ε, στόχων του ορίζοντα Ευρώπης και σε όλο το πρόγραμμα. Δεύτερο σημείο οι κοινωνίες που θα είναι ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί. Θα ήταν καλό αν μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό και για, τους, για το φάκελο Ορίζον Ευρώπη και για το ειδικό πρόγραμμα. Καλωσορίζουμε το κλάστερ για την ψηφιακή βιομηχανία. Θα πρέπει όμως να εστιαστούμε περισσότερο στο κλίμα και στην ενέργεια. Αν σκεφτούμε ότι η βιομηχανία ε, είναι ε, αυτή που παράγει τις Υψηλότερε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Σα ευχαριστώ. Χωρί μικρόφωνο η πρόεδρο. Yeah. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω για την έκθεση του συνέφου του Ντανίκα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παραγωγή συνεργασία που επιδιώκει να έχει με όλε τι πολιτικέ ομάδε, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ομάδα της GUNGL βλέπει εν γέννη θετικά τις πρώτες προτάσεις που καταθέσει ο εισηγητής για την έκθεση Horizon Europe. Σίγουρα συμφωνούμε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ορθή ισορροπία μεταξύ της συνέχισης της ανοιχτής επιστήμης και καινοτομίας και της διασφάλισης των επιστημονικών και οικονομικών συμφερόντων της κοινωνίας και των λαών της Ένωσης. Η ερευνητική ατζέντα θα πρέπει να διαμορφωθεί δίνοντας προτεραιότητα στα προγράμματα που ανταποκρίνονται πραγματικά σε σύγχρονε ανάγκε τη κοινωνία και κατά νέα όψη μα όχι σε αυτά που ξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Έτσι μόνο θα υπάρξουν πραγματικά κοινωνικά ωφέλη. Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγηση, έχοντα τώρα και την εμπειρία του προγράμματο Ορίζοντα 2020, θα πρέπει να επιδιώξουμε βελτιώσει, μεγαλύτερη διαφάνεια και δίκαια διαμορφωμένε ομάδε αξιολόγηση με εκπροσώπους από όλα τα κράτη-μέλη. Ε, στόχος είναι να πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες που υπήρχαν μέχρι σήμερα όσον αφορά την πρόσβαση των χωρών στη χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στη συμμετοχή των τρίτων χωρών ώστε να αποφευχθούν κρούσματα που υπήρξαν στο παρελθόν όπου μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται φορείς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τέλο είναι σημαντικό να επισημάνουμε ε, πω τα δεδομένα και οι γνώσεις που θα παράγονται από τα έργα, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Όση, πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα διαμορφώσουμε και τι δικέ μα τροπολογίε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ματίας, που είναι σκιώδης για το ειδικό πρόγραμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα κάνω κάποια γενικά σχόλια στο στάδιο αυτό. Συμφωνώ με πολλά πόσα υπόθηκαν. Απλώς να αναφερθώ σε κάποιες ανησυχίες που έχω. Είτε ως προς το περιεχόμενο, είτε προς το θέμα της οργάνωσης. Χρειάζονται κάποιες διευκρίνισεις πιστεύω, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος αυτό καθ' αυτό. Με ανησυχεί το θέμα της σύγκληση και της συμπερίληψης ε, στον πυλώνα της ε, βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας με τις παγκόσμιες προκλήσεις. Κυρίως όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη αποσαφήνιση για το ποιο είναι το ποσό της ε, κάθε βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και για κάθε παγκόσμια πρόκληση. Και αν αυτό δεν γίνει, υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος να ε, αφαιρέσουμε από την επιστήμη ε, και από την κοινοτομία βασικούς πόρους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη διάκριση και αυτή την αποσαφήνιση και να εγγυηθούμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε σχέση με τις παγκόσμιες προκλήσεις, ε, κάτι που αφορά το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Θα ήθελα και σαφή διάκριση εντός του δεύτερου πυλώνα αυτό που έχουμε για τις ασφαλείς ε, κοινωνίες και χωρίς διακρίσεις. Είχαμε την ίδια συζήτηση και στον ορίζοντα 2020 και πετύχαμε ε, κάτι και ελπίζω να διατηρηθεί και εδώ. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες ε, είναι θεμελιώδη εργαλεία. Εμείς δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στις κοινωνίες, πάνω σε κοινωνίες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να εγγυθούμε να έχουμε αυτόνομη χρηματοδότηση για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είμαι ικανοποιημένοι με το ότι αυξάνεται ο προπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, όμω θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι θα είναι απόλυτα αυτόνομο το Συμβούλιο αυτό. Έχω ε, κάποιες ε, ε, αμφιβολίες σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των κόλ, τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι αυτό θέτει κάποιο βάρος μεγαλύτερο στους ερευνητές και στα πανεπιστήμια και επίσης ε, υπάρχει και το θέμα της ε, ίσης αμοιβή για ισότιμη εργασία. Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με τα εργαλεία για το στρατηγικό συνδυασμό. Δεν υπάρχει καμία σαφήνεια. Ε, εδώ μιλάμε για πιλωτικά σχέδια ή για κάποιες συμπράξει. Πρέπει να δούμε και ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν ορίζεται σαφώς η αυτονομία, το ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και με ανησυχεί και η μείωση των κονδυλίων για τι υποδομέ. Ευχαριστώ. Εκτό μικροφώνου, πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση ο συνάδελφος Νίκα γιατί ποτέ δεν είχα μέχρι τώρα δει κάποιον που ξεπέρασε τις πολιτικές του πεπιθήσεις και συνεργάστηκα με τόσο καλά. Νομίζω πως πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ε, σίγουρα, ε, αυτό το σχεδιάζουμε κιόλα. ένας λοιπόν ε, διαχωρισμός από, του, από την χωρίς αποκλεισμούς από τη μία και από τη δημιουργική κοινότητα. Αυτό ήταν κάτι που μας απασχολούσε πάντα. Και πάντα υπήρχαν φόβοι πως ε, το ένα θα επηρεάσει αρνητικά τον προϋπολογισμό του άλλου. Νομίζω πως ε, θα έπρεπε να δώσουμε στο Συμβούλιο και την Κομισιόν κάποια ελευθερία έτσι ώστε να ε, δώσουν ε, ορισμούς. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση πρέπει να είναι αυτό που θα προτιμήσουμε. Χρειάζεται όμως να μην ε, ξεχνάμε πως ε, πρέπει να δούμε το θέμα με τις αποστολές εξίσου γρήγορα, διότι δεν είναι ε, απλά αρκετό να τελειώνουμε και να αφήνουμε δύο χρόνια το θέμα με τις αποστολές. Έπειτα, τα διάφορα επιμέρους προγράμματα για την αριστεία, για την προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή. Έχετε δίκιο μετά η ενιαία προσέγγιση με βάση τον δημοσιονομικό κανονισμό είναι πολύ σημαντική. Με, σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς μας, ε, το 60% των σφαλμάτων προέρχεται από αυτούς τους τομείς. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Η ταχεία προσέγγιση πρέπει να διευρυνθεί σε περισσότερους τομείς. και ο περιορισμός των καταποκοπή ποσών χωρίς προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις θα έπρεπε να ε, περιέχουν τουλάχιστον μία αξιολόγηση, κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει στην διάμεση αξιολόγηση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ε, διευρύνουμε έτσι απλά αυτά τα πόσα χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες και πώς ακριβώς ε, επηρεάζουν τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ. Εμείς πρέπει να πούμε στον αυτό μας την αλήθεια. Αυτές οι δύο εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης. Και η πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, όπως και ο κανονισμός για, τον ορίζον, για το ορίζον Ευρώπη. οι συνάδελφοι προσπάθησαν να ακούσουν ώστε να τον περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να προσπαθήσουν να ε, παρουσιάσουν μία πρόταση όσο το δυνατόν λιγότερο αποδεκτή. Μία πρόταση ε, που θα πρέπει να αντικατοπτριστεί με πολύ μεγάλη προσοχή και στο ειδικό πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Θα πρέπει να εργαστούμε ε, και στους δύο φακέλους σε πολύ στενό χρονικό διάστημα και φυσικά αυτό υποσκάπτει την ποιότητα της δουλειάς μας και μάλιστα αποφασίστηκε να ακολουθηθεί μια ατζέντα που ζητήθηκε από την Κομισιόν που ε, τελικά είναι εις βάρος ε, τη συμμετοχή των stakeholders αλλά και εις βάρος της δικής μας συνεισφοράς. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι εκούσια επιλέχθηκε η ταχύτητα έναντι της ποιότητας για να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος ε, της ε, θητείας. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι κάποιοι βουλευτές ε, σκέφτηκαν να συνεισφέρουν στην, επιτυχ... στην επιτάχυνση της διαδικασίας προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα για τις επόμενες ευρωεκλογές. Έτσι λοιπόν, καθώς πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα για το μέλλον, δεν θα ήταν ε, καλύτερο ε, να αναβληθεί ε, μία εργασία, γιατί θα έπρεπε να διέπεται από ποιότητα και διαφάνεια η νομοθεσία αυτή. Έτσι λοιπόν, θα ήταν καλό να μεταφέρουμε εντό του κανονισμού όλα τα νομοθετήματα. Θα είχαμε ένα και μόνο κανονισμό που διαφύλασε τις αρμοδιότητές μας ε, και χωρίς να έχουμε γκρίζες ε, ζώνες. Έτσι λοιπόν θα ασχολείται με όλες ε, τις πτυχές και με το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού. Τώρα για να μπούμε στην ουσία. Θα ήθελα να πω ότι ο συμπληρωματικό προπολογισμό δεν είναι ικανοποιητικό. Αντίθετα, το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων θα ήταν πιο ικανοποιητικό για του τομεί ε, αυτού του τομέα. Υπογραμμίζω ότι η κατανομή του προπολογισμού μεταξύ διάφορων πυλώνων και για τα διάφορα κλάστερ ε, του ε, πυλώνα βιομηχανική ανταγωνιστικότητα παγκόσμιε προκλήσεις ε, μας δημιουργεί προβλήματα επίσης και για τις ασφαλείς κοινωνίες και για τους τομείς του κλίματος και της κινητικότητας υπάρχει μείωση του προπολογισμού σε σχέση με το σημερινό ορίζοντα 2020 επίσης θεωρώ ότι το κείμενο ευνοεί την βιομηχανία των αγορών και Επομένως, ε, τελικά δεν σέβεται την έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές αοριστείες, όπως ε, οι αποστολές, παραδείγματος χάρη. Η Κομισιόν θα μπορεί να κάνει τον πραγματικό στρατηγικό σχεδιασμό, είναι όμω πολύ σημαντική η διαδικασία της συναπόφασης, όπως ορίζεται και στις συνθήκες. Και σημειώνω με πικρία ότι εξαφανίστηκε το μέσο για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Λείπει ε, ο κατάλληλος τρομές του υπολογισμού για αυτές. Σε σχέση με τις εταιρικέ σχέσεις έχουμε τρεις διαφορετικές ε, τυπολογίε ομαδοποίηση με ιδιώτε. Όμως νομίζω ότι δεν έχουμε εδώ τη δυνατότητα σχέση σχέσης δημοσίου-δημοσίου. Είμαι κάπως διστακτική και στις επιχειρήσεις με χρηματοδότηση, χρηματοδότησης, blending, που θελοποιηθούν με το Ταμείο InvestEU. Ε, εδώ θα ήταν απαραίτητο να εισαχθούν μηχανισμοί για να αποφύγουμε ότι να έχουμε τυχαίες ε, οικονομικές ε, πράξεις έτσι ώστε να ε, μπορούν να βασιστούν στην πραγματική οικονομία οι συμμετέχοντες. Εγώ από την πλευρά μου μετά από όλα αυτά θέλω να προσφέρω και την πλήρη συνεργασία μου για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτό θα πάρω και εγώ, λέει η Πρόεδρος, για να επαναλάβω μια έννοια που ήδη εκφράστηκε στην εξαιρετική έκθεση του κυρίου Ντανίκα αλλά νομίζω την ανέφερε και ο κύριος Έλερ και η Καμπεσόν Ρουίς, αλλά και άλλοι. Και κόβεται το μικρόφωνο της Πρόεδρου. Το θέμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που όπως είπα επαναλήφθηκε από όλου. Θα ήθελα και η Κομισιόν να, να ακούσει αυτή την ισχυρή φωνή που ακούστηκε από εμά Πολύ ωραία όλα αυτά που μας έχετε βάλει στον πυλώνα της καινοτομίας και της ικανότητας στο βιομηχανικό μας σύστημα να είναι πιο ανταγωνιστικό χάρη και στην ε, παρέμβαση και στη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας κυρίως στην Ευρώπη. Όμως, σε αυτό το ποιοτικό άλμα που είναι τόσο σημαντικό, δεν μπορούμε να ξεχνάμε και το εργαλείο, το μέσο για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, το Fast Track, που είχε τόσα πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, ε, υπήρχαν τόσα πολλά project, όμως ε, λόγω έλλειψης πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τις χώρες μας. Όλοι γνωρίζουμε μικρές πραγματικότητες που ακόμη και με περιορισμένες καινοτομίες, κάποιο προϊόντος ίσως, εγώ έχω κατά νου μια επιχείρηση στην περιοχή μου, που άλλαξε τη σύνθεση, το χάρη της ε, ύλης ασφαλτόστρωσης, της πίσας, χάρη σε αυτή την αλλαγή που οφείλεται στην ε, έρευνα για να έχουμε ένα προϊόν ε, πιο βιώσιμο, αυξήθηκε η δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν ήταν μια καινοτομία προβληματική, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική γενοτομία. Θα ήθελα να σας πω και άλλα, αλλά σας ακούσαμε και για το θέμα της υγείας, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα ήθελα η Κομισιόν να καταλάβει ότι η δική μας Επιτροπή ανησυχεί πάρα πολύ για αυτό το μέσο που δεν το βλέπουμε πλέον μήπω θα μπορούσε να υπάρχει μια δυνατότητα και για αυτή την καινοτομία που μπορεί να συνεισφέρει στο γενικό καλό. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Μαντερβίβε, που τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει τους συζητητές ε, που παρουσίασαν σήμερα τα βασικά χαρακτηριστικά των ε, σχεδίων έκθεσης. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να επενθυμίσουμε τα λόγια του Επιτρόπου, γιατί όταν ήρθε στην Επιτροπή πριν από ένα περίπου μήνα είπε ότι σήμερα έχουμε μία μοναδική ευκαιρία και το ίδιο ισχύει και κατά τους επόμενους εβδομάδες και μήνες να αναδιαμορφώσουμε την καινοτομία προς το καλύτερο. Προσβλέπουμε λοιπόν στο να υπάρχει ένας καλός ε, σχεδιασμός από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, σημειώσαμε αυτά που είπα για τον προπολογισμό, αυτό που προτείνεται, ο προπολογισμό των 100 δις ευρώ είναι η αναγνώριση της πολύ σκληρής δουλειάς που έγινε για την αναγνώριση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και είναι και ψήφος εμπιστοσύνης από την Επίτροπο Γιούνκερ που σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό γίνονται επενδύσει για το μέλλον της Ευρώπης. Χαιρετίζουμε πολλές από τις προτάσεις που ακούσαμε σήμερα από τις ηγητές μοιάζουν να στηρίζουν τη δική μας την πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα να γίνει σχεδιασμός κατά το μέγιστο Αυτά που ακούσαμε σήμερα έχουν ως στόχο να κινητροδοτήσουν τη συζήτηση ακούσαμε τις ανησυχίες σας που έχουν σχέση με, τον, ε, με τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτός, πιο διαφανής σε σχέση με αυτά που ισχύουν τώρα ε, στην ε, διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού υπό το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο τρόπο μαζί σας κατά τις επόμενες εβδομάδες. Επιπλέον, ε, χαιρετίζουμε το ότι πολλοί ομιλητές μίλησαν για το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα, όχι μόνο ανάμεσα στα διερθωτικά ταμεία, αλλά και με το πρόγραμμα Erasmus και Creating Europe. Ενδεικτικά τα λέω αυτά. Επίσης, καταγράψαμε και τις προκλήσεις όπου πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές κυρίως για να περιοριστεί το χάσμα καινοτομία στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία που θα καταλήξει σε νέες φιλοδοξίες στον τομέα της έρευνα και καινοτομίας. Όπως είπε και ο Επίτροπος πριν από ένα μήνα εδώ, είμαι πεπισμένος ότι με το πρόγραμμα Horizon Europe μπορούμε να να επιφέρουμε ουσιαστική διαφορά. Και έτσι η Κομισιόν συμμερίζεται την επιθυμία του ε, Κοινοβουλίου να ολοκληρωθούν το συντομότερο διαπραγματεύσεις υπό το σύνθημα ποιότητα και ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω την Προεδρία στον Πρόεδρο Μπούζεκ. Νομίζω ότι σήμερα το πρωί, για σήμερα το πρωί αξίζεται τις ευχαριστίες μας ε, γιατί σας εκτιμούμε για το πώ χειριστήκατε την ε, ψηφοφορία το πρωί. Ευχαριστώ, Πατρίτσια. Αφού βγήκα από αυτή την αίθουσα, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Τώρα όλα είναι καλά. Well, ή uh, uh, μισή ώρε ε, πέρασαν και έπινα νερό συνεχώς. Είναι επικίνδυνο αυτό, πρέπει να προσέχετε. Λοιπόν, οι συγητές μας. Ο κύριος Ντανίκα και ο κύριος Έλερ. Έχουν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, από τους σκιώδεις εισηγητές και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Λοιπόν, έχουμε πάνω κάτω 15 λεπτά και θα προσπαθήσω να δώσω μία κατάλληλη απάντηση στις διάφορες ανησυχίες που υπάρχουν και ορθώς τέθηκαν από όλους τους πήραν το λόγο. Μία κυρία ανησυχία υπάρχει και για μένα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα 120 δισεκατομμύρια πραγματικά θα δοθούν στους ερευνητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα. Και σε συνεργασία με άλλα ε, αξιόλογα Ινστιτούτα στον κόσμο θα υπάρξει προκειμένου να εξελιχθούν και τα εμπόδια για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια προκειμένου η αρχή της αριστείας ε, να είναι αυτή που επικρατεί όχι να έχουμε να υπερισχύουν κριτήρια φύλου ή γεωγραφικά κριτήρια και για να είναι οι εμπειρογνώμονες ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες όλες αυτές ε, τις ανησυχίες προσπάθησα και εγώ να τις ε, απαντήσω στην έκθεση μάλιστα θα ήθελα και η κοινότητα των Ευρωπαίων Ερευνητών να λάβει μια κατάλληλη απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια, αξιοπιστία και πολύ καλύτερη κατανόηση του πώς γίνεται η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η πρόσβαση θα πρέπει να γίνεται με ένα και μόνο στόχο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει η έρευνα να ωφελεί τους Ευρωπαίους πολίτες καθώς είναι αυτοί που πληρώνουν για αυτή την ερευνητική δραστηριότητα. Και να επαναλάβω το εξή από τα 100 ευρώ που δίνονται σε δαπάνες για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 7 ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ τα 93 από εθνικά κονδύλια. τα ευρωπαϊκά κονδύλια μάλλον όσοι ε, αναφέρθηκαν στα ευρωπαϊκά κονδύλια παρακαλώ να το ψάξουν ε, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα να χρησιμοποιούνται τα εθνικά κονδύλια γιατί τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι αρκετά χαμηλά ε, σε σχέση με τις τεράστιες ε, ανάγκες και τα τεράστια αιτήματα που υπάρχουν από τους ευρωπαίους ερευνητέ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο κύριος Θα ήθελα ε, να αναφερθώ στα κρίσιμα ερωτήματα που ετέθησαν. Πράγματι πρόκειται για ένα ε, φιλόδοξο πρόγραμμα, όπως είπε και ο Επίτροπος, είναι θαραλέο, αναφέρεται στις ε, προκλήσεις ε, παγκόσμιου βεληνικούς που αντιμετωπίζουμε. Ε, Παραδείγματο χάρη, ποια είναι η βάση τη ευημερία στην Ευρώπη. Η ευημερία ανέκαθεν βασιζόταν στην ικανότητά μα για καινοτομία. Ζούμε πλέον σε ένα τελείω διαφορετικό κόσμο. Λόγω τη ψηφιοποίηση, λόγω τη ε, ταχύτητα και νομίζω ότι πλέον έχει προσθεθεί και ένας νέος πυλώνας που δίνει πάρα πολλές απαντήσεις. Θέλω όμως να πω και το εξής, ότι όσον αφορά το σύνθημα ταχύτητα υπέρ τη ε, ποιότητα, Αυτό δεν ισχύει. Ε, συστήσαμε μία ομάδα εργασία ε, και θέλουμε να εξετάσουμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η πρόταση της Κομισιόν. Το δεύτερο που θέλω να πω την ταχύτητα δεν την θεωρούμε ως ιδέα, αλλά στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα τα οποία ξεκινάνε σιγά σιγά τα πρώτα δύο χρόνια, τα τελευταία εξελίσσονται, εκτινάσσονται θα έλεγα και μετά ξαναπέφτουν. Αυτό όμως δεν αντιστοιχεί ούτε στη συνέχεια, ούτε στην ασφάλεια, ούτε στην ανταγωνιστικότητα που θέλουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι που είναι οι ερευνητές, τα πανεπιστήμια και η βιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρέπει να προτιμούμε απαραίτητα την ταχύτητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δίνουμε απαντήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι και στην καινοτομία βοηθάει τους ανθρώπους να είναι κανείς ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι στην αιχμή του δόρατος όσον αφορά τις εξελίξεις. Και θέλουμε ταχύτητα, γιατί στην περίπτωση αυτή θα έχουμε το προνόμιο ότι αν του χρόνου ολοκληρώσουμε τότε η κοινωνία θα μπορεί να βασίζεται σε αυτόν τον κύκλο των δύο ετών για νέα προγράμματα, για ε, ομίλους επιχειρήσεων. Θέλουμε την κβαντοπληροφορική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια νύχτα. Η κβαντοπληροφορική δεν μπορεί να υπάρχει ήδη τον Ιανουάριο του 2021. Ήδη τώρα πρέπει να δώσουμε τα σημαντικά μηνύματα. Θέλουμε κβαντοπληροφορική υπολογιστική. Ε, θέλουμε νέα κλάστερ. Ε, θέλουμε καινοτομία. Ως εκ τούτου η ταχύτητα δεν είναι η προσπάθεια να τα συγκαλύψουμε. Είναι αυτό που πρέπει πραγματικά να κάνουμε, δηλαδή οφείλουμε να ε, ανταπεξέλθουμε, να μετρηθούμε με το ε, παγκόσμιο, την παγκόσμια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η μόνη που είναι αργή δεν είναι οι ερευνητές, ούτε επιχειρηματίες, ούτε πανεπιστημία αργή. είμαστε εμείς. Αν για 18 ολόκληρους μήνες δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα. Ε, να πούμε έχουμε 120 δις, έχουμε φιλοδοξίες, θέλουμε να, να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι να προηγείται η ταχύτητα της ποιότητας, αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αν θέλουμε ή έχω απαιτήσει έναντι των ερευνητών, των επιχειρηματιών και των πανεπιστημίων, ε, τότε πια και εμείς θα πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε έναν στόχο. Όχι αδιαφανή. Και δεν είναι βλακεία ότι δεν δίνουμε εξουσιοδότηση εν λευκό. Ε, αναφέρεται ότι η Κομισιόν ε, και το Συμβούλιο θέλουν κάποια εξουσιοδότηση. Όχι, εμείς θέλουμε εξουσιοδότηση πράξη. Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ, να μην το ε, διατυμπανίσετε αυτό στην κοινή γνώμη, ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι η ταχύτητα έναντι της ποιότητας. Όχι, αυτό που ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα και το μήνυμα προς τους επιστήμονες ότι και εμείς μπορούμε να είμαστε ταχύτεροι αν τελικά μεταβάλλονται συνθήκες συνεχώς ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ε, νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική συζήτηση λίγο πριν ε, από τις ε, διακοπές και ας μην ξεχνάμε, είχαμε τέσσερις υπουργούς από την Αυστριακή Προεδρία σήμερα το απόγευμα και μια καταπληκτική συζήτηση για το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon τελειώσαμε μεγαλοπρεπώς θα έλεγα ως Επιτροπή Ήτρε και θα ήθελα να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στις 3 ε, και στις 24 Σεπτεμβρίου, δύο Δευτέρες είναι αυτές, το απόγευμα και τα δύο απογεύματα θα έχουμε συναντήσει της Επιτροπής Ήτρε με ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν να είστε έτοιμοι 4 ώρα το απόγευμα, στις 3 και στις 24 Σεπτεμβρίου. Επίσης, ενδεχομένως να έχουμε μια συνάντηση και στις 18 Σεπτεμβρίου. Είναι πράσινη εβδομάδα και πολλές πολιτικές ομάδες, οι περισσότεροι, ε, διαμαρτυρήθηκαν γιατί είπαν όταν είναι πράσινη εβδομάδα δεν είναι καλό να συνεδριάσει η Επιτροπή Ήτρε. Εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουμε από αυτού και μπορούμε να ακυρώσουμε αυτή την συνεδρία. Και θέλω να σας πω ότι αν είναι απαραίτητο Μια επιπρόσθετη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο στις 10 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, τη νύχτα ή το απόγευμα, βράδυ, δεν ξέρω ίσως ε, από τις 7 μέχρι τις 10 και μισή. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι για επιπρόσθετη συνεδρία της Επιτροπής Ήτρε στο Στρασβούργο στις 10 Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα ε, στις 3 και στις 24 όπως είχε προβλεφθεί. Καλές διακοπές. Ξεκουραστείτε γιατί οι επόμενες διακοπές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα είναι τελείως διαφορετικές. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών και για τις δύο εκθέσεις 6 Σεπτεμβρίου του 18. Όλες οι τροπολογίες και για τις δύο εκθέσεις. Καλές διακοπές φίλοι μου, γεια σας.